και στη συνέχεια θα ακούσουμε και τους κοιόδους συγγητές βέβαια που θα σχολιάσουν συντομία. Η κάτι πύρη έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση για την Τελωνιακή Ένωση και την γνωμοδότηση να πω μια φράση. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 11 ε, αντιφρονούντες οι οποίοι βρίσκονται στη φυλακή και οι βουλευτές είναι στη φυλακή και πρόσφατα συνελήφθησαν και άλλοι. Ε, έχουν παγώσει προσωρινά οι διαπραγματεύσει με την Τουρκία ακριβώς επειδή οποιαδήποτε κριτική φωνή αυτή τη στιγμή διώκεται. Είτε είναι ακαδημαϊκή, είτε είναι πολιτική, είτε είναι δημοσιογράφη. Ξέρουμε ότι ο πολιτικός διάλογος είναι πολύ τεταμένος με την Τουρκία λόγω της κατάστασης αυτής και ακολουθούμε λοιπόν παρόλα αυτά όμως να θέτουμε τα ζητήματα αυτά στο διάλογο με την Άγκυρα. Σε αυτό το πλαίσιο η Ευρωπαϊκή η Επιτροπή θα ζητήσει από το Συμβούλιο επίσημη εντολή ε, για να ξεκινήσει εξχρονισμός της Τελωνιακής ε, Ένωσης ε, που ορίζει και τη σχέση μας με την Τουρκία. Η Τελωνιακή Ένωση ήταν υποφελής και για τους δύο. Η Τουρκία είναι ο έκτος εμπορικός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο πρώτος για την Τουρκία. Είναι όντως πεπαλαιωμένη αυτή η Τελωνιακή Ένωση, πρέπει να εξχρονιστεί ε, πρέπει να διευρύνει το πεδίο της, το πεδίο της αυτό, αυτή την αρχή την υποστηρίζει η Επιτροπή μας εδώ και χρόνια. Βεβαίως έχουμε πολιτικές διαφορές όταν συζητούμε το κατά πόσο πρέπει η Τουρκία να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμφωνούμε όμως όλοι ότι κάποια μορφή συνεργασίας πρέπει να υπάρχει. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η ίντα θέλει να επηρεάσει ε, την εντολή δίνοντας την ε, άποψή τη πριν ξεκινήσει τι διαπραγματεύσει. Εμεί έχουμε γνώμη μόνο για, το, για την έκθεση πρωτοβουλία. Έχουμε πει όμω στον ενδιάμεσο εισηγητή ότι δεν θα ήταν σοφό να βιαστούμε με την έκθεση αυτή στο Ευρωκοινοβούλιο λόγω του ευαίσθητου του ζητήματο. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα του timing, διότι αυτή τη στιγμή εξακολουθούμε να έχουμε καθώ έκθεση ανάγκη στην Τουρκία. Ε, τρία ζητήματα αναφέρουμε εμεί στην έκθεσή μα. Καταρχήν, ο εξοχρονισμό τη Ελληνική Ένωση θα κρατήσει την Τουρκία ε, οικονομικά ε, δεμένη με την Ευρώπη και αυτό είναι καλό. Βεβαίως οι μεγάλες γεωπολιτικές και οικονομικές ε, προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τουρκικός λαός είναι κάτι που πρέπει να μας υποσχολήσει. Ναι, οι κανόνες λοιπόν είναι σημαντικοί και έτσι τις τουρκικές επιχειρήσεις έτσι ώστε το περιβαλλοντικό για ε, το επιχειρηματικό περιβάλλον να είναι πιο σταθερό, αλλά και για, και για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Και τέλος, και ίσως και σημαντικότερο, εμείς να γνωρίζουμε ότι αυτές οι διαπραγματεύσεις μπορούν να διαρκέσουν πολλά χρόνια, ε, είναι όμως σημαντικό να συμπεριλάβουμε, παρότι μιλάμε για μια εμπορική σχέση, να συμπεριλάβουμε και κάποια πολιτικά benchmarks σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως έχουμε κάνει στο παρελθόν ε, στις πιο πρόσφατες ε, εμπορικές συμφωνίες με τρίτες χώρες. Αυτά είχα να πω εγώ πρόεδρε και βεβαίως αναμένω να ακούσω και την άποψη των σχεδόν συγκητών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Κατυπέρη. Η Σκιώδης. Η Ζώμα από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι γεγονό ο εξυγχρονισμό τη Τελωνική Ένωση είναι απαραίτητο. Γνωρίζουμε ότι είναι πεπαλαιωμένο ε, το νομικό πλαίσιο και θα πρέπει να διευρυνθεί ακριβώ έτσι ώστε η Τουρκία να συνεχίσει να είναι δεμένη με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τι οικονομικέ μα σχέσει. Και υπάρχει δυνατότητα επέκταση ε, στη γεωργία, στι υπηρεσίε, στι δημόσιε συμβάσει ενδεχομένω τη Τελωνιακή Ένωση. Ε, και είναι και αμοιβαία αποφελής αυτός ε, ο εξχρονισμός. Υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν θα πρέπει να λησμονούμε. Θυμίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην τρέχουσα ετήσια έκθεση διαπιστώνει ότι πέρυσι δεν ε, επετεύχθη πρόοδος καθόλου στην Τελωνιακή Ένωση τα διάφορα μέτρα για τη ζώνη ελευθερών συναλλαγών και η διαχείριση των ποσοστώσεων δεν συνάδει απολύτως με το κοινοτικό κεκτημένο ούτε με τις συμβατικές υποχρεώσεις της Τουρκίας και εν μέρει οι κανόνες παραβιάζονται κιόλας και αυτά είναι γνωστά. Επίσης και επιπλέον το τελωνιακό δίκαιο θα πρέπει να εναρμονιστεί με τον Ευρωπαϊκό Τελωνιακό Κώδικα. Και διερωτώ με, μήπως μπορούμε να κάνουμε κι εμείς τροπολογίες στη δική μας επιτροπή. Αυτό θα το κρίνει ο πρόεδρος, αν είναι παραδεκτές ή όχι οι τροπολογίες μας. Αλλά γνωρίζουμε ότι η Τουρκία εδώ και καιρό ε, έχει κάποια ελλείμματα που πρέπει να καλύψει εκτός από την Τελωνιακή Ένωση και κάτι που είναι δική μας αρμοδιότητα στην Επιτροπή μας, η Τελωνιακή Ένωση μπορεί να αξιοποιηθεί πλήρως μόνο εφόσον η Τουρκία ε, ε, εφαρμόσει πλήρως το συμπροματικό πρωτόκολλο έναντι όλων των κρατών μελών μας και θα πρέπει να το λέμε αυτό έξω από τα δόντια. Το λέει και κάτι πύρη. Ο εξυγχρονισμός είναι κι άλλος ένας μοχλός για μας έτσι ώστε να πιέσουμε την Τουρκία και να της ασκήσουμε επιρροή. Θυμίζω ότι ε, στο τελευταίο μας ψήφισμα του Νοεμβρίου του 2016 διαπιστώσαμε ότι έχει ε, μεγάλες οικονομικές επιπτώσεις ενδεχομένως και για την Τουρκία ε, η καθυστέρηση και η κατάργηση αυτών των προσπαθειών και αυτό θα πρέπει να το θέτουμε υπόψη της Τουρκίας. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Φροντίστε τις τροπολογίες σας να τις κάνετε στην Επιτροπή Ίντα, αν θέλετε να είναι παραδεκτές. Και μην αρχίσουμε τώρα αυτή τη διελκυστίδα ε, για τις αρμοδιότητες. Ε, μας είπε Ίντα ότι εκεί πρέπει να πάνε οι τροπολογίες. του Τζέφρι Βαν Όρντεν. Ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ πάντα υπήρξα υπέρ των ε, ορθολογικών σχέσεων, ρεαλιστικών σχέσεων με την ε, Τουρκία. Ε, και βεβαίως εδώ πρέπει να δούμε κατά πόσον θέλουμε να ενθαρρύνουμε την Τουρκία να έρθει πιο κοντά μας ή αν θέλουμε να την απομακρύνουμε άλλο περισσότερο, ακόμη περισσότερο. Ε, πρέπει να πω ότι η δουλειά της Κατυπήρη γενικά είναι πολύ καλή, πολύ σωστή και έχει πάρει μια πολύ λογική προσέγγιση. Αλλά υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία θα ήθελα να αναφέρω. Ας πούμε στην παράγραφο 1, παρότι ε, θέλουμε η Τουρκία να παραμείνει οικονομικά κοντά ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είμαι βέβαιος ότι χρειάζεται να το πούμε εξπρέσεις verbis νομίζω ότι θα πρέπει να μην το λέμε τόσο ρητά και να κάνουμε έτσι μια πιο και καλυμμένη διατύπωση. Ε, τελευταία φράση στην παράγραφο 1 όπου κάνετε αναφορά ε, στην ε, ε, θετική, στο θεωτικό θεματολόγιο, μετριάζοντας ταυτόχρονα και την πολιτική κατάσταση. Νομίζω ότι εκεί μπορείτε να το σταματήσετε. Δεν υπάρχει λόγος να αναφέρετε την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών στη χώρα. Γνωρίζουμε πώς είναι η κατάσταση, δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να την αναφέρουμε ρητά εδώ. Στην παράγραφο 5 Δεν είμαι βέβαιος ότι μπορεί κανείς να εξάγει το συμπέρασμα που έχετε εξάγει βάσει ε, της ε, Ένωσης, ε, της Τελωνιακής Ένωσης. Νομίζω ότι είναι σαφές ότι είναι καλό για την Τουρκία να έχει Τελωνιακή Ένωση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα το κατά πόσον αυτό την έχει κάνει πιο αναπτυγμένη, αυτό είναι διαφορετικό και πιο ανταγωνιστική. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα συμπέρασμα που δεν ε, είναι αυτόματο. Ε, κοιτάξτε, σε όρους οικονομικής ε, ανάπτυξης το μοντέλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι πράγματι ένα μοντέλο το οποίο θέλουμε να ακολουθήσουν και άλλοι. Είναι υπερβολική λοιπόν αυτή η διαπίστωση στην παράγραφο 5. Αυτές είναι οι παρατηρήσεις μου για την ώρα. Ε, αλλά σε γενικές γραμμές ε, βεβαίως ε, μπορώ να, να στηρίξω την εργασία σας. Ο κύριος Κατζηγεωργίου, επόμενος Κιώδης. Καλημέρα σε όλους σας. Εγώ εδώ βλέπω μία προσπάθεια να κρατηθεί η Τουρκία σε τροχιά γύρω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί κανείς βεβαίως ε, να κατανοήσει το γιατί της θέσης αυτής. Ωστόσο, εγώ πιστεύω ότι εμείς έχουμε παγιωθεί στο παρελθόν, σε διαδικασίες που είχαν ακολουθηθεί στο παρελθόν και που κατά την άποψή μου είναι πλέον πεπαλαιωμένες και επομένως δεν λειτουργούν ούτε σήμερα ούτε θα λειτουργήσουν και θα έχουν αποτέλεσμα αύριο. Πιστεύω ότι πρέπει ριζικά να τροποποιήσουμε τη θέση μας απέναντι στην Τουρκία όσο κρατάει η Τουρκία κλειστά τα λιμάνια της ε, ε, για ε, πλοία ή αεροπλάνα που έρχονται από την Κύπρο, όσο δεν εφαρμόζει την υφιστάμενη τελωνιακή ένωση απέναντι στην Κυπριακή Δημοκρατία, τότε πιστεύω ότι είναι σαφές σε όλους μας ότι εάν δεν λυθούν τα ζητήματα αυτά και εάν δεν εφαρμοστούν πλήρως, τότε δεν είναι δυνατόν να εξυγχρονιστεί η υφιστάμενη τελωνιακή ένωση. Δεν θέλω να διευρύνω περισσότερο το θέμα, ωστόσο πιστεύω ότι οικονομικά ζητήματα πάντα τα οικονομικά ζητήματα έχουν και κάποια σχέση με την δημοκρατία. Και δεν είναι δυνατόν να λησμονούμε τα όσα συμβαίνουν τούτη τη στιγμή στην Τουρκία. Και σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να στείλουμε σε αυτή τη χώρα ε, οποιοδήποτε θετικό μήνυμα, να κάνουμε οποιαδήποτε θετική χειρονομία. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, δεν βλέπω άλλους σκιώδεις συγητές που να θέλουν να πάρουν το λόγο, επομένως μπορούμε να συνεχίσουμε με άλλα ε, μέλη. Ο κύριος Βίστεσεν, from, from... αντιπρόεδρος. Από πλευράς ε, της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων νομίζω ότι σημαντικό είναι να δούμε την πλήρη εικόνα της ε, Τουρκίας, να δούμε και την Τουρκία και σαν υποψήφια χώρα ε, και σαν χώρα που έχει ειδικέ σχέσεις και λόγω ΝΑΤΟ και τα λοιπά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σημαντικό πάντως, πολύ σημαντικό, ε, στις συστάσεις σας, στη σύσταση 6, να γίνει λόγος για το benchmark και για την δημοκρατία. Μιλάμε για τη σχέση μας με την Τουρκία σε μια στιγμή όπου πολλά πράγματα πηγαίνουν στη λάθος κατεύθυνση και όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και όσον αφορά δημοκρατικές αρχές και όσον αφορά την ανεξάρτη, τις ανεξάρτητες δικαστικές αρχές. Ε, και δεν πρέπει να λησμονούμε ότι η Τουρκία είναι και υποψήφια χώρα και επομένως οτιδήποτε κάνουν προς αυτήν έχει κάποιο βάρος. Δεν είναι δυνατόν να δίνουμε κάτι από τη μία και να παίρνουμε κάτι ε, από την ε, άλλη. Θα πρέπει να δούμε ε, βεβαίως τα θετικά στοιχεία των εμπορικών συναλλαγών αλλά μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σαλή από την Άλτε. Ευχαριστώ πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι. Καταρχάς, θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Πύρη για το σχέδιο γνωμοδότησης της που υπογραμμίζει ε, ε, τη σημασία του εξυγχρονισμού της Τελωνιακής Ένωσης και την αμοιβαία επωφελής αυτή η προσπάθεια. Όπως ε, περιγράφει, εμείς οι Ευρωπαίοι εταίροι της Τουρκίας υποστηρίζουμε κάθε θετική εξέλιξη που είναι αμοιβαίως επωφελής και για τις δύο πλευρές σήμερα και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τουρκία αντιμετωπίζουν κοινά προβλήματα ε, αρχίζει γενομένης από την οικονομική κρίση μέχρι τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Είναι κρίσιμη εταιρική σχέση μα από πλευρά οικονομικών σχέσεων. Είναι ο πέμπτο μεγαλύτερο εμπορικό μα εταίρο. ενώ εμείς είμαστε παριθμόν ένα για την Τουρκία. Εξού και η σημασία για την Τελωνιακή Ένωση και η επιθυμία μα να βελτιώσουμε τη λειτουργία τη. Δεν χωρά καμία αμφιβολία ότι είναι πάρα πολύ σκόπιμο να διαβρεθεί και να εξυγχρονιστεί η Τελωνική Ένωση για να ρυθμίσουμε τις διμερείς μας σχέσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει την Τουρκία στις συνεννοήσεις για τις διεθνείς συμφωνίες ε, όπου μετέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι δημόσιες υπηρεσίες, ε, η γεωργία και οι δημόσιες συμβάσεις είναι θέματα που κυριαρχούν στις συζητήσεις μας και θα πρέπει να εκτιμήσουμε, ε, να δούμε ποιο θα είναι το πραγματικό πεδίο εφαρμογή της διεύρυνσης Τελωνικής Ένωσης. Και τέλος, ο εξυγχρονισμός της Τελωνικής Ένωσης θα είναι ένα κοινό βήμα ενδεχομένω για τη βελτίωση των σχέσεων μας παρά τις μεταβαλλόμενες συνθήκες, ο διάλογο υψηλού επίπεδου θα πρέπει να συνεχίσει να διευρύνεται και να εμβαθύνεται. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ. Ο κύριος Σολέ. Εκ μέρου των Πρασίνων, ε, η Τουρκία για μια σειρά από λόγου είναι στρατηγικό εταίρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η οικονομική συνεργασία είναι σημαντική, για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ταυτόχρονα υπάρχει μια αύξηση στην ένταση και στην περιπλοκότητα του εμπορίου τα τελευταία χρόνια. Οπότε η παρούσα Τελωνιακή Ένωση θα πρέπει να βελτιωθεί ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαπραγματεύσεις οι ενταξιακές έχουν παγώσει και δεν υπάρχει κάποια προοπτική να ξεκινήσουν εκ νέου. Βεβαίως η επιδείνωση του κράτους δικαίου και των θεμελιών δικαιωμάτων στη χώρα αυτή, καθώς και ενσχυτική κατάσταση ε, στο τουρκικό Κουρδιστάν, καθώς και το θέμα των προσφύγων, είναι ζητήματα που μας απασχολούν ιδιαίτερα, μας ανησυχούν. Ε, δεν είναι λοιπόν κατά τη γνώμη μας η κατάλληλη στιγμή να ξεκινήσουν οι πραγματεύσεις ε, για την επικαιροποίηση της Τελωνιακής Ένωσης τώρα όταν βλέπουμε την Τουρκία να ακολουθεί το δρόμο των ανελευθεριών και, του περιορισμού του κράτους δικαίου. Δεν είναι τώρα η στιγμή ε, του εξχρονισμού της Θελωνιακής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Σακουράφα έχει το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώντας την κυρία Πύρη, πρέπει να πω πρώτα και πάνω απ' όλα ότι μια πιθανή αναβάθμιση της παροχημένης Θελωνιακής Ένωσης που βρίσκεται σε ισχύ για περισσότερα από 21 χρόνια θα πρέπει να σέβεται καταρχήν τις ιδιαιτερότητες που υπάρχουν στην, και τις ευαισθησίες που υπάρχουν στην περιοχή. Και το λέω αυτό γιατί καλούμαστε να τοποθετηθούμε σαν Επιτροπή για το συγκεκριμένο ζήτημα σε μια περίοδο που ο κύριος Ερντογάν εξασφαλίζει την παντοδυναμία του πάνω στη δυστυχία των προσφύγων, πάνω στα συντρίνια της δημοκρατίας, με μαζικές εκαθαρίσεις στη δημόσια διοίκηση και με συλλήψεις και κατηγορίες για εθνική προδοσία Κούρδων πολιτών και πολιτικών. Με απειλέ προ τι γειτονικέ χώρε, με παραβιάσει αναέριων και θαλάσσιων συνόρων τη Ευρωπαϊκή Ένωση και φυσικά με την αμφισβήτηση του στάτου quo τη περιοχή. Συμφωνώ απόλυτα με την εισηγήτρια ότι υπάρχει ανάγκη για μια τέτοια αναβάθμιση, αν φυσικά καταλήξει κάποτε να εμπεριέχει σαφεί ρήτρε προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που δεν θα αποτελούν απλά διακοσμητικό στοιχείο, όπω συμβαίνει για πολλέ από τι συμφωνίε που έχει υπογράψει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τρίτε χώρε. Επιπλέον, είναι ανάγκη να συσταθεί ένα σύγχρονο αυτόματο δεσμευτικό μηχανισμό επίλυση διαφορών, ώστε να εκλείψουν οι συμπεριφορέ παραβιάσεων τη Τελωτινιακή Ένωση που παρατηρήθηκαν από την τουρκική πλευρά όλο το προηγούμενο διάστημα. Τέλο, κύριοι συνάδελφοι, καμία αναβάθμιση δεν μπορεί να εφαρμοστεί αν η Τουρκία δεν συμμορφωθεί με τι ευρωπαϊκέ υποχρεώσει για την πλήρη εφαρμογή του πρόσθετου πρωτοκόλλου προ όλα τα κράτη-μέλη και την αναγνώριση φυσικά τη Κυπριακή Δημοκρατία. Ευχαριστώ. Thank you, Next is Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Σχάκε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ζητή συγγνώμη ο κύριος Λάμστροφ ε, για την απουσία του. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Κάτι για το σχέδιο γνωμοδότησης. Είναι καλό και είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε αυτή τη διπλή προσέγγιση που θέλουμε και επιζητούμε. Έχει δίκιο το Κοινοβούλιο όταν τονίζει τη σημασία του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτου δικαίου ε, στην Τουρκία και ζητούμε πάγωμα των προενταξιακών διαπραγματεύσεων. Πέρα από αυτό όμω, παράλληλα, έχουμε το θέμα τη ε, ενημέρωση και επικαιροποίηση τη Τελωνιακή Ένωση. Είναι, όπω ακούσαμε, πεπαλαιωμένη πρώτον. Η ιδέα τη Τελωνιακή Ένωση ήταν ότι ήταν ένα πρώτο βήμα προ την πλήρη ένταξη. Τώρα βλέπουμε ότι δεν προβλέπεται αυτό ε, στο στο άμεσο μέλλον από κανέναν. Άρα υπάρχει ανάγκη ουσιαστική να αναβαθμιστεί και να εξυγχρονιστεί η τρέχουσα τελωνιακή ένωση. Δεν σημαίνει αυτό ότι δεν έχουμε ευκαιρίες να εντάξουμε και τις αρχές ε, στη συζήτηση και να πούμε ότι είναι αναπόσπαστο στο τμήμα ε, της πολιτικής μας και της εμπορικής. Πάντα μας ενδιαφέρει αυτό. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ε, τα benchmarks που θέλουμε στην ε, ενημέρωση της Ελληνικής Ένωσης, στον εξυγχρονισμό της και πάντα ε, σε ό,τι κάνουμε κυριαρχούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και άλλο πράγμα είναι να αρχίσει τη συζήτηση για τον εξοχρονισμό και άλλο να την τελειώσει. Δεν σημαίνει ότι τελειώνει εδώ αυτή η υπόθεση ε, για την έναρξη τέτοιων συζητήσεων. Δεν θέλουμε να κόψουμε όλου του δεσμού και τι σχέσει που έχουμε με την Τουρκία. Ευχαριστώ. Τρεις τελευταίους ομιλητές έχουμε. Τον κύριο Λόπες, τον κύριο Μπέλτερ και τον κύριο Επιτίδιο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομος. Θέλω να υποστηρίξω το προσχέδιο της συναδέλφου μου ε, Κατυπήρη, κυρίως γιατί πιστεύω ότι πρέπει να κρατήσουμε ανοιχτή την προοπτική με την Τουρκία ε, και επίσης λαμβάνοντας υπόψη και τα μηνύματα που έχουμε στείλει τον τελευταίο καιρό. Πρώτον, ότι δηλαδή θα πρέπει η Τουρκία να παραμείνει συνδεδεμένη με την ε, Ευρώπη και βεβαίως ε, ε, ε, ε, λαμβάνοντας υπόψη το πολιτικό πλαίσιο και εκεί να στείλουμε πολύ αυστηρά μηνύματα τα οποία σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις παραβιάσεις παντός είδου στην Τουρκία. Επομένως πρέπει να υπάρξει η, η, ο εξυγχρονισμός αυτός αλλά να υπάρξουν ρήτρε πολύ συγκεκριμένε για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε αυτή τη χώρα, όπως ακριβώς είπε ε, και η συνάδελφο Κάτι Πύρη. Ευχαριστώ, Μπασμπέντερ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Το κόμμα μου ε, αναγνωρίζει ε, τα όσα λέει η Κάτι Πύρη και ξέρει ότι εμείς ε, έχουμε πάντα συνεπή στάση ως κόμμα απέναντι στην Τουρκία. Δεν θέλουμε να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θέλουμε ε, ανέκαθεν να εμβαθυνθεί η τελωνιακή ε, ένωση. Αλλά είναι οι πολιτικές εξελίξεις τόσο δραματικές αυτή τη στιγμή στην Τουρκία με διώξεις δημοσιογράφων και το Φόρουμ Ανεξαρτήτων Δημοσιογράφων ε, στη Γερμανία το καταγγέλει και το βρίσκω πάρα πολύ προβληματικό αυτή τη στιγμή να προωθούμε τέτοια διεύρυνση ε, της Θελωνιακής Ένωσης. Και αν δούμε την τελευταία παράγραφο ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις ε, ελευθερίες, πόρο απέχει από όλα αυτά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει ξεδοντιαστεί το Κοινοβούλιο, έχει αποδυναμωθεί το λίος είναι πάρα πολύ προβληματικό για την επόμενη περίοδο να συζητάμε τέτοια πράγματα και ακόμα και για τον εξυγχρονισμό της Τελωνιακή Ένωσης. Ευχαριστώ. Τελευταίος ομιλητής ο κύριος Επιτήδιος. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η θέση ότι ο εξυγχρονισμός της Τελωνιακή Ένωσης ε, με την Τουρκία θα φέρει πιο κοντά την Τουρκία ε, είτε ότι θα μπορέσει να αποτελέσει μοχλό πιέσεως της Ευρωπαϊκή Ένωσης προς αυτήν είναι περισσότερο ένας ευσεβής πόθος και λιγότερο μια πραγματιστική αντιμετώπιση της καταστάσεως. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η Τουρκία δεν σέβεται τις συμφωνίες τις οποίες συνάπτει και πάντοτε ενεργεί σύμφωνα με το συμφέρον της, χωρίς βεβαίως να διστάζει να εκβιάζει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι δυνατόν η Τουρκία να μην αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία, να μην επιτρέπει την πρόσβαση των πλοίων και των αεροσκαφών της Κύπρου στους λιμένες και τους αρελιμένες της και εμείς θα συζητούμε εδώ για αναβάθμιση των εμπορικών σχέσεων με την Τουρκία. Άλλωστε αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν επήγει να συμβεί. Και επιπλέον το να δίνουμε δώρα στην Τουρκία δεν σημαίνει ότι θα την κάνουμε πιο διαλλακτική και συνεργάσιμη. Αντιθέτως, θα την κάνουμε περισσότερο προκλητική και θα την αποθρασύνουμε. Ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστώ. Για τα καταλεκτικά σχόλια, δεν ξέρω αν θέλει η συντάκτρια της νομοδότησης να πει κάτι. Κάτι πήρε σύντομα, λέει κυρία Πύρη. Καταρχάς, ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τη σημαντική του συνεισφορά και από την πολύτιμη. Ε, να αρχίσω από εκεί που σταμάτησε η Μαρίκε Σχάκε. Αυτή είναι έκθεση πρωτοβουλίας ε, του Κοινοβουλίου και εμείς νομοδοτούμε απλώς και μόνο είτε γνωμοδοτήσουμε είτε όχι ως κοινοβούλιο, το Συμβούλιο ξέρετε ότι μάλλον θα δώσει εντολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αρχίσει διαπραγματεύσεις. Οπότε είναι πολύ χρήσιμο να πει κάτι το Κοινοβούλιο, να δώσει τη γνώμη του, να πει πώς βλέπει τη διαδικασία. Βεβαίω, μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων που μπορεί να χρειαστούν και δύο και τρία χρόνια, είναι μακρά πνοή, η ενδεχόμενη συμφωνία θα επανέλθει στο Κοινοβούλιο για τη σύμφωνη γνώμη του. Και τότε θα είναι η στιγμή να πούμε ε, τι φρονούμε υπό το φω των τότε πολιτικών εξελίξεων και άλλων. Αλλά τώρα θα ήταν μια χαμένη ευκαιρία να μην ακούσει η φωνή του Κοινοβουλίου ε, για τι διαπραγματεύσει αυτέ. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Κύπρο, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και ε, ο εισηγητής στην ίντα και παρακαλώ διαβάστε την έκθεση ίντα, το έχουν ξεκαθαρίσει. Μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η συμφωνία θα πρέπει να εφαρμόζεται και για τα 28 κράτη-μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου. Βεβαίω το Κοινοβούλιο συμφωνεί με αυτό. Και ένα τελευταίο σχόλιο προς εκείνους και τον Αντίπρόεδρο της Επιτροπής μας που ε, ε, μαζευστούν την προσοχή στα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες. Το Κοινοβούλιο μας ήταν το μόνο θεσμικό όργανο όπου έχει με τις υποψήφιες χώρες και συγκεκριμένα με την Τουρκία ε, πολύ ψηλά στις προτεραιότητες στα ανθρώπινα δικαιώματα ε, και τις θεμελιώδεις ελευθερίες. Δεν πρόκειται να καταργηθούν αυτά από τη συγκεκριμένη γνωμοδότηση. Αλλά ακόμα και αν δεν μπούμε τίποτα. Ακόμα και δεν συζητούμε για την ένταξη της Τουρκίας. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Είναι ε, και σημαντικό η χώρα για μας και στρατηγικός εταίρος. Κάποιο είδους συνεργασία πρέπει να έχουμε με την Τουρκία. Οικονομικά είμαστε άρρηκτα συνδεδεμένοι. Ας μεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία να έχουμε περισσότερους κανόνες γιατί το ζητούν οι επιχειρήσεις και μάλιστα και οι τουρκικές επιχειρήσεις ε, επικρίνουν οξύτατα τη σημερινή κατάσταση. Να αξιοποιήσουμε αυτό το μοχλό που έχουμε βεβαίω για την ενταξιακή διαδικασία διαδικασία το Κοινοβούλιο εξακολουθεί να το βλέπει με πάρα πολύ κριτική ματιά. Γι' αυτό το λόγο, Πρόεδρε, σας μίλησα για, για τους 12 και όχι 11 συναδέλφους βουλευτές που κρατούνται αυτή τη στιγμή, βουλευτές της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης. Θα τα συζητήσουμε αυτά ξανά και με τους υπόλοιπους και οδησίγητες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Κάτι Πύρη, συντάκτες νομοδότησης. Και τώρα μπορούμε να ολοκληρώσουμε αυτή την κυκλισμένη των θυρών συνεδρίαση. 1η ε, Φεβρουαρίου, αύριο 6 η ώρα το απόγευμα, λίγη προθεσμία για τις τροπολογίες, ενώ στις 28 Φεβρουαρίου το πρωί θα ψηφίσουμε εδώ στην Επιτροπή μας. Και πάμε στο επόμενο θέμα, που είναι δημόσια ακρόαση. Ο Nord Stream 2 και για πολιτικές του συνέπειες. Έχετε λάβει ένα χωριστό πρόγραμμα για την ακρόαση αυτή. Θέλω να καλωσορίσω όλους ε, τους συμμετέχοντες σε αυτή την πολύ επίκαιρη συζήτηση ε, για το έργο αυτό και τις γεωπολιτικές προεκτάσεις. Ξέρω ότι έχει γεννήσει πολύ ενδιαφέρον και σε μερικούς ε, ανησυχίες και σε κάποια κράτη-μέλη μας. Οι ανησυχίε βεβαίως είναι ποικίλε, νομικές, γεωπολιτικέ, οικονομικές, περιβαλλοντικές. Πολλοί από εσά τι ε, αναφέρατε και το Μάιο και το Νοέμβριο ε, σε σχέση με την πολιτική ενεργειακή ασφάλεια της Ένωσης. Βεβαίως όλα τα ενεργειακά μας έργα θα πρέπει ε, να συνάδουν με τους στόχους μας και της ασφάλεια και του ενεργειακού ενεφοδιασμού. Ε, θεωρώ πολύ σημαντικό να το συζητούμε αυτό το θέμα ε, στην Επιτροπή μας γιατί το θέμα της ενεργειακής ασφάλειας είναι πολύ σημαντικό στην εξωτερική μας δράση και ε, συχνά τα συζητούμε αυτά τα θέματα από το πρίσμα της ασφάλειας. Από την αρχή του έργου αυτού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Διαστόματος Εύκοβιτς, Κανιέτε και Γιούνκε μίλησε για κίνδυνο ε, μεγαλύτερης εξάρτησης ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Ρωσία εάν ε, ε, κατασκευαστεί ο αγωγός Nord Stream 2 θα αλλάξει το πεδίο και η εικόνα προμήθειας φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Πολωνική Αρχή Ανταγωνισμού εκφράζει μερικές ε, και σοβαρέ επιφυλάξει. Ορισμένοι Ευρωπαίοι ε, εταίροι έχουν αποσυρθεί και η Gazprom ε, κυριαρχεί. Εδώ καλέσαμε σήμερα λοιπόν τρεις εμπειρογνώμονες εγνωσμένου κύρους για να μας παρουσιάσουν τις απόψει του. Είναι ο κύριο Ανδρέας Κόλταου, καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Royal Holloway του Λονδίνου και επίσης συμμετέχει και στο Πανεπιστήμιο ε, του Χάρβαρτ, στο Belfer Center για την επιστήμη και τις διεθνείς ε, ε, υποθέσεις και σε ένα ρωσικό Ινστιτούτο. Έχουμε τον κύριο Σέμπρεν Ντε Γιόγκ, στρατηγικό αναλυτή στο κέντρο της Χάγης Στρατηγικών Σπουδών και στο Λάινταν διδάσκει, έχει διδακτορικό στην ε, σχέση εξωτερικής ασφάλειας από το Πανεπιστήμιο της Λέβαν και έχει και σπουδάσει οικονομική γεωγραφία στο Πανεπιστήμιο του Χρόνιγκεν. Και έχουμε και τη κυρία Στραχώτα ε, που είναι ερευνήτρια στο στη Βαρσοβία, ε, στο Κέντρο Ανατολικών Σπουδών ε, και ερευνά θέματα ενεργειακής πολιτικής, αγοράς φυσικού αερίου και τη διάσταση κυρίως της εξωτερικής ασφάλειας, σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας ε, στο φυσικό αέριο και επιπτώσεις για την Ανατολική Ευρώπη. Καλώς ορίζω και τους τρεις εμπειρογνώμονες, θέλω να τους δώσω το λόγο και ως προς το χρόνο έχουμε προγραμματίσει να ε, θα τους ακούσουμε μέχρι τις 11.30 και από τις 11.30 μέχρι τις 12 και 4 να ακολουθήσει συζήτηση. Ε, και το αργότερο στις 12.30 θα τελειώσει η πρωινή συνεδρίαση. Έχουμε 50 λεπτά λοιπόν για τις ε, παρουσιάσεις. Ο καθένας σας μπορεί να μιλήσει 15 λεπτά. Ποιος θέλει να ξεκινήσει.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 Ελάτε εδώ να μιλήσετε. Εδώ στο Προεδρείο. Ε, ίσως είναι καλύτερα. Μόνο φιλικά πρόσωπα θα δείτε. Και εσείς, και εσείς οι δύο, ελάτε από τώρα βεβαίως. Ναι, ελάτε, ελάτε στο Προεδρείο. Έχει καλύτερη θέα, επαναλαμβάνω. Λοιπόν, έχετε το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Είναι μεγάλη τιμή για μένα που συμμετέχω σε αυτήν την πολύ σημαντική επιτροπή και να μιλήσω μάλιστα και εδώ, στο Πρόεδρο του Νέου, θα λέω στην τηλεόραση αυτά. Τώρα είμαι στην τηλεόραση. Είναι λοιπόν τιμή και χαρά που είμαι εδώ μαζί σας. Θα ήθελα ποιος, να ρωτήσω ποιος από εσά θεωρεί ότι το Nord Stream δεν είναι καλή συμφωνία. Ποιο θεωρεί ότι δεν είναι καλή συμφωνία, ότι είναι κακή συμφωνία για την Ευρώπη. Ωραία. Ποιο από εσά θεωρεί ότι αυτό έχει να κάνει με οικονομικά στοιχεία, ότι είναι οικονομικό το πρόβλημα. Και ποιο θεωρεί ότι είναι για πολιτικούς λόγους κακό. Ωραία. Λοιπόν, φαίνεται να μην λειτουργεί αυτό. Μια στιγμούλα. Μπορείτε να με βοηθήσετε. Ναι. Οι απόψεις εδώ, σε αυτή την αίθουσα και στην Επιτροπή, ουσιαστικά αποτυπώνει και τις απόψεις της διαπραγματεύσης γενικότερα. Ο Τζο Μπάιντεν είπε ότι το Nord Stream 2 είναι κακή ε, επιλογή για την Ευρώπη. Συγγνώμη. Όπως είπε και ο Πρόεδρος, ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στους Ευρωπαϊκούς Αξιωματούχους ε, λέγεται ότι θα μειωθεί η ασφάλεια λόγω του Nord Stream 2, ε, γίνεται αναφορά στις γεωπολιτικές επιπτώσεις και επιπλέον έχουν υποθεί πολλά, έχουν γίνει συζητήσεις και για το νομικό σκέλος του ζητήματος και σε ποιο βαθμό η ευρωπαϊκή ενεργειακή νομοθεσία θα εφαρμιστεί στο Nord Stream 2 και κατά πόσο ο Nord Stream 2 τελικά υπόκειται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ε, εμένα μου ζητήθηκε να μιλήσω για το οικονομικό σκέλος, αλλά ε, θα αναφερθώ λίγο και στο νομικό. Τα γεωπολιτικά θα τα αναφέρει θα τα οι θα τα αναφέρουν οι συνάδελφοι εδώ στο πάνελ. Πρέπει να διευκρινίσουμε όμω πρώτα περί πρόκειται. Ξέρω ότι είστε εξοικειωμένοι με τον Nord Stream 2 γενικότερα μιλάμε ε, για έναν αγωγό 55 PCM που θα έρθει να υποκαταστήσει έναν άλλον αγωγό θα οδηγήσει σε 110 PCM ε, ε φυσικού αερίου προς την Ευρώπη στη Γερμανία που είναι η μεγαλύτερη αγορά στην ε, ε Ήπειρο είναι 90 PCM η αγορά δηλαδή καλύπτει τη Βαλτική, την Πολωνία και τη Γερμανία μόνο αυτός ο αγωγός. Η Gazprom τον έχτισε, τον δημιούργησε από το 2016 ε, με τη σύμπραξη κάποιων ευρωπαϊκών εταιριών. Αυτό βεβαίως άλλαξε διότι οι πολωνικές αρχές έβαλαν βέτο ε, σε αυτήν την σύμπραξη και τώρα η Gazprom προχωράει μόνη της, λέει ότι θα προχωρήσει και το project προχωράει έγκαιρα, είναι εντός χρονοδιάγραμματος δηλαδή, εάν δούμε τουλάχιστον αυτά που λένε οι Ρώσοι. Τώρα, τι σημαίνει ε, για την αγορά και την αγορά αερίου πιο συγκεκριμένα το Nord Stream 2. Για να καταλάβουμε αυτό, καλό θα ήταν να δούμε τι έκανε το Nord Stream 1 ε, που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η αγορά φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Εδώ βλέπετε τις ροές φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Τις ροές λοιπόν από τη Δύση προς την Ανατολή, πηγαίνοντας προς τα κάτω, ε, κάτω έχουμε την Ουκρανία ε, και, και έχετε και το καφέ την καφέ γραμμή που πάει προς τα πάνω που είναι το Nord Stream, το Nord Stream. Δηλαδή το Nord Stream μείωσε τις ροές φυσικού αερίου από την Ουκρανία. Αυτό άλλωστε είχε σκοπό να κάνει η Gazprom ε, και αυτό γίνεται και με τον Nord Stream 2, ίσως και περισσότερο. Η ιδέα λοιπόν είναι ε, να εργαστούμε χωρίς την Ουκρανία ως χώρα transit. Όμως υπάρχει και ένα δεύτερο στοιχείο που παρουσιάζει ενδιαφέρον εδώ. Όταν το Nord Stream έφτασε στην υπηρετική Ευρώπη, στην ε, Βαλτική θάλασσα, στη Γερμανία, άρχισε να, ανταγωνίζεται ε, το φυσικό αέριο από την Νορβηγία, το, υγρό, το υγραέριο ε, και αυτό σε ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό περιβάλλον λόγω και κάποιων νομοθετικών πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως το τρίτο πακέτο ενέργειας του 2009. Έτσι λοιπόν η Γκάσπρο μάχησε να ανταγωνίζεται με άλλες πηγές αερίου και άρχισε να ξεπερνάει το αέριο ε, που προερχόταν από την Ουκρανία. Και αυτό που βλέπετε εδώ στο γράφημα είναι ότι ξαφνικά η Τσεχία, η Σλοβακία, ακόμα και η Ουκρανία άρχισαν να παίρνουν ε, φυσικό αέριο από τη Δύση και από την Ανατολή, γιατί ήταν ευθυνότερο. Είναι λοιπόν αρκετά ηρωνικό ε, Ρώσοι ανταγωνίζονται Ρώσους, Ρώσοι από τη Δύση ανταγωνίζονται Ρώσους από την Ανατολή. Ε, απλώς ήταν πιο φτηνά, τα αγόρασαν οι έμποροι καταναλωτές στη Δυτική Ευρώπη και, αυτό το, και σε αυτό βοήθησαν οι υποδομές. Οι υποδομές που βοήθησαν στη διασύνδεση των εθνικών ε, αγορών αερίου έχουμε πολλά δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ε, τα οποία περνάνε από αυτές τις υποδομές. Ένα άλλο στοιχείο είναι ότι οι ανατολικές, ε, οι αγορές άρχισαν να ε, ενσωματώνονται, να συνδέονται με δυτικούς ε, θύλακες, δυτικούς κόμβους μάλλον ενέργειας ο συνάδελφός μου, ένας συνάδελφός μου τον έφερε αυτό ε, ο, ο νόμος ε, των ε, μη επιδιακόμενων επιπτώσεων. Άλλαξε λοιπόν ο τρόπος με τον οποίο γίνεται, ε, λειτουργεί αγορά αερίου στην Ευρώπη. Κάτι ακόμα. Δεν είναι μόνο, ότι, δεν είναι μόνο ανταγωνισμός μεταξύ διαφόρων πηγών φυσικού αερίου, αλλά υπάρχει πλέον η δυνατότητα, η εναλλακτική να βρει κανείς φθηνότερο φυσικό αέριο από τη Δύση. Ε, εδώ βλέπετε τις διασυνοριακές τιμές εισαγωγής ε, για το αέριο από, το, από τη Ρωσία που φτάνει στην Ανατολική Ευρώπη σε σχέση με τις τιμές στα, σύνορα ε, της Γερμανίας. Εδώ βλέπετε ότι αυτές τις τιμές άρχισαν σιγά σιγά να συγκλίνουν και στη συνέχεια να πέφτουν. Στην ε, νοτιοανατολική Ευρώπη υπήρξε η δυνατότητα να έρχονται λοιπόν, έχει το αέριο φτηνότερο από τη Δύση και έτσι οι ανατολικές χώρες αναδιαπραγματεύθηκαν τις συμφωνίες με τη Ρωσία. Και αυτό ήταν υπέρ του καταναλωτή. Θα ήθελα να αναφερθώ τώρα στο νομικό σκέλος του συστήματος, ότι περνάει ο χρόνος. Εδώ βλέπετε ένα τόμο που είναι η ενεργειακή νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι κάτι που συζητείται εδώ και καιρό και για τον Nord Stream 2, για το ρωσικό φυσικό αέριο και γενικότερα για την αγορά φυσικού αερίου της Ένωσης. Το ζήτημα λοιπόν είναι σε ποιο βαθμό το Nord Stream 2 υπόκειται στην νομοθεσία αυτή και στου νομικού διακανονισμούς που έχουν προκύψει με μια σειρά από ενεργειακά πακέτα από το δεκαετία 1990 και μετά. Εάν παρακολουθήσετε τις δημόσιε, συζητήσει, τη δημόσια συζήτηση, ε, λέγεται ότι η Gazprom και όσοι εν πάση μπαίνουν στην αγορά την Ευρωπαϊκή πρέπει να σέβονται τους κανόνες της Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ δεν συμφωνώ απόλυτα. Δεν είναι τόσο απλό το Nord Stream 2 είναι ένας αγωγός offshore. Δεν καλύπτεται από το ενεργειακό καθεστώς της Ένωσης. Καλύπτεται από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του ε, Δικαίου της Θάλασσας, την UNCLOS. Υπάρχουν βεβαίως συμφωνίες διακυβερνητικές που καλύπτουν αυτές τις πτυχές των αγωγών και τα συστήματα ασφάλειας, ε, συντήρησης, ε, ε, ανωτέρα βία κτλ. Γι' αυτό λοιπόν κανεί, κανείς από εισαγωγής από τη Μεσόγειο, από την Αλγερία, από τη Λιβύη δεν υπόκεινται στο ενεργειακό καθεστώς της Ένωσης. Από την Νορβηγία ναι, αλλά η Νορβηγία είναι μέλος του Ευρωπαϊκού, Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Είναι δύσκολο λοιπόν να πει κανεί να πείσει με επιχειρήματα ότι η Nord Stream 2 πρέπει να υπόκειται στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Εάν θέλετε να το κάνετε αυτό, τότε πρέπει να που απαντήσετε στο εξή ερώτημα. Για ποιον αγωγό μιλάμε. Μιλάμε για έναν αγωγό διασύνδεσης. Σύμφωνα με το άρθρο 34 του Νεγιακού πακέτου, είναι ένας αγωγός που συνδέει δύο αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ισχύει αυτό. Η Ρωσία είναι μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ή μιλάμε για έναν αγωγό upstream που φέρνει, φέρνει αέριο στην ευρωπαϊκή αγορά. Τότε υπάρχει πρόβλημα. Διότι αυτή η αγωγή εξαιρούνται από τις προϋποθέσεις του τρίτου ενεργειακού πακέτου και πρέπει να πιστοποιηθούν από τη χώρα ε, όπου φτάνει ο αγωγός, δηλαδή στην προηγούμενη περίπτωση στη Γερμανία. Είναι δύσκολο λοιπόν να πει κανείς ότι το Nord Stream 2 πρέπει να υπόκειται στο καθεστώς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν θέλετε να το κάνετε, τότε θα πρέπει να εξηγήσετε ότι το Nord Stream συνδέει αγορές της Ένωσης Λέει βέβαια, λένε κάποιοι ότι περνάει από τη Δανία, περνάει από τη Σουηδία, όπω περνάει από τη Γερμανία, περνάει από διάφορε ζώνε ευρωπαϊκέ. Αλλά αυτό κατ' εμέ ε, είναι αρκετά σε επιχείρημα. Τώρα, χρειάζονται οι επεκτάσεις onshore. Το Nord Stream 1 φτάνει στην Κλάισφαρτ στη Γερμανία, προέρχεται από την ΟΠΑΛ, ε, ένα αγώνα που μπορείτε να έχετε παρακολουθήσει και έχουν γίνει πολλές συζητήσεις γι' αυτό, νομικές, όσοι έχουν τα πράγματα 5% ε, καλύπτεται η χρήση του ε, υπήρξαν κάποιες συμφωνίες το 2016 το Δεκέμβριο μεταξύ Γκάσπρομ και Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι το Gazprom, η Gazprom μπορεί να προβεί σε όποιες αλλαγές θέλει. Δεν θέλω να σας κουράσω με τις, ε, ε λεπτομέρειες. Ε, κάποιοι ήταν κατά, τώρα το θέμα έχει πάει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ε, η ΟΠΑΛ, δεν χρησιμοποιείται και το Nord Stream 1 δεν χρησιμοποιείται πλήρως λόγω αυτού του γεγονότος. Βεβαίως η Gazprom έμαθε μετά από 8 χρόνια ε, συζητήσεων για την ΟΠΑΛ και το Nord Stream 2 δεν θα είναι ΟΠΑΛ, δεν θα είναι ούτε ΟΠΑΛ θα είναι ένα διαφορετικός αγωγός και θα ακολουθεί ένα διαφορετικό καθεστώς. Θα έχουμε έναν αγωγό που ε, θα ε, το διοικεί ένας ανεξάρτητος ε, πιστοποιημένος ε, επιχειρηματίας. Εάν διαβάσετε το τρίτο ενεργειακό πακέτο και αυτά που λέει, είναι πιθανό αυτός ο αγωγός να συμμορφώνεται με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Βεβαίως η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία δεν είναι πάντα απολύτως συμπαγής, πάντα αφήνει κάποια περιθώρια ερμηνείας, Υπάρχει όμω κάτι το οποίο είναι κάπω επικίνδυνο εάν αρχίσουμε, να παίζουμε πολύ με τι ερμηνείε ε, της νομοθεσίας. Ιδιαίτερα αν την εφαρμόζουμε επιλεκτικά, διότι ουσιαστικά πολιτικοποιούμε του κανόνε, ε, οι κανόνε υπάρχουν για να λειτουργεί η αγορά και ιδιαίτερα σε αφορά την ενεργειακή αγορά θέλουμε να έχουμε ίσες ευκαιρίε για όποιον ε, μπαίνει στην ευρωπαϊκή αγορά. Αν αρχίζουμε τώρα να λέμε ότι υπάρχουν καλοί και κακοί, αυτό γίνεται. Αλλά ε, θα μπαίνετε εδώ σε έδαφο Τραμπ, για να το πω έτσι. Λέμε αυτά είναι καλά αυτοκίνητα, αυτά είναι κακά αυτοκίνητα, θέλουμε αυτά, δεν θέλουμε τα άλλα. Δεν πρέπει να κάνει τέτοια πράγματα ένα κανόνα νομικό. Διότι αυτό πολιτικοποιεί τη ρυθμιστική αρχή, που είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και πολιτικοποιεί τον ίδιο τον κανονισμό. Έχω ακόμα ένα λεπτό. Ε, και να φτάσω στο θέμα της Ουκρανίας, ε, που είναι σημαντικό το θέμα αυτό στην συζήτηση. Πολλά ελέγχθησαν για τα δύο δισεκατομμύρια που θα χάσει η Ουκρανία ε, σε, έσοδα λόγω του Nord Stream 2. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά κάποια στιγμή εξετάσα και τα στοιχεία ε, σε σχέση με την ε, αποζημίωση που έλαβε η Ουκρανία, μάλλον την έκπτωση το 2014, το 15 και το 16. Εδώ βλέπετε το, τι έγινε το 15 τις εκπτώσεις. εάν τα συγκρίνετε αυτά και το πολλαπλασιάστε με τα 16 BCM που λαμβάνει από τη Ρωσία η Κουρανία, τελικά έχουμε 1,1 δισεκατομμύρια σε 100 ε, κέρδη. Ε, δεν θα καλύψει βέβαια 3 δισεκατομμύρια ε, ε, απολειών, αλλά κάποια χρήματα που είναι στα ε, δημόσια ταμεία θα βρεθούν στα, στις τσέπες των καταναλωτών και των επιχειρήσεων. Ε, και αυτό για μια χώρα που έχει προβλήματα οικονομικά και που δυσκολεύεται να σταθεί στα πόδια της, ίσως να μην είναι και τόσο κακό. Κλείνοντας, τέσσερα σημεία. Πρώτον, θεωρώ ότι το Nord Stream 2 μπορεί από οικονομικής πλευράς και από νομικής πλευράς ε, από οικονομικής πλευράς, περιπτώσει, να μην, μπορεί να μην είναι τόσο προβληματικό. Βεβαίω υπάρχει το πολιτικό σκέλο, έτσι. Αλλά για τον καταναλωτή υπάρχει κέρδο. Η προπόθεση γι' αυτό είναι να υπάρχει κάποιο ισχυρό επόπτη σε επίπεδο, σε επίπεδο ανταγωνισμού. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. χρειάζεται ε, interconnectors, στοιχεία διασύνδεση. Θα το δούμε και αυτό. Είναι σημαντικό η εκλεκτική πάντως και στρατηγική χρήση της νομοθεσίας δεν είναι καλή ιδέα, δεν πρέπει να το κάνει κανείς αυτό. Εάν το ρωσικό φυσικό αέριο αμφισβητείται για λόγους ασφάλειας, είναι κάτι που πρέπει να εξεταστεί. Ε, δεν είναι κάτι το οποίο θέλω να αποφύγω συζήτηση, αλλά εάν αμφισβητείται για λόγους ασφάλειας, τότε πρέπει αυτό να εξεταστεί σε, επίπεδο πολιτικής, ε, όχι σε επίπεδο τεχνικό, οικονομικό, το οποίο όμως πολιτικοποιούμε. Αυτά, Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Thank you, Mr. Uh, for Ευχαριστώ κύριε Γκόλταου για την πρώτη αυτή παρουσίαση. Επόμενος εμπειρογνώμων που θα λάβει το λόγο, ο κύριος Σίμπρεν Ντεγιόγκ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση που μου απευθύνεται για να μιλήσω στην Επιτροπή σας. Τρία πράγματα θέλω να τονίσω. Πρώτον, ο βαθμός στον οποίο το έργο Nord Stream 2 μπορεί να θεωρηθεί εμπορικό έργο, γιατί υπάρχουν πολλά θέματα γεωπολιτικά και ασφαλείας που θα αναλύσω στη συνέχεια και θα ήθελα να τελειώσω ε, ευρύτερα ε, γεωστρατηγικά θέματα ε, που αφορούν και άλλους αγωγούς όπως τον τουρκικό. Τα θέματα ανταγωνισμού τα είπε ο συνάδελφος Γκόλταου. Από πλευράς επιχειρηματικής είναι αξιοσημείωτο που φαίνεται κάθε φορά να υπερεπενδύουμε σε αγωγούς για ορυκτά καύσιμα. Ε, όχι μόνο μειώνεται αυτή τη στιγμή η ζήτηση για το φυσικό αέριο και αυξάνεται για το υγροποιημένο αέριο, αλλά και γιατί είναι εκπεφρασμένο στόχο μακροπρόθεσμα να γίνουν επενδύσει σε ανανεώσιμες ε, πηγές ενέργειας και σε καθαρή ενέργεια. Τούτου λεχθέντος υπάρχει και απόφαση ε, της Πολωνικής Αρχής Ανταγωνισμού και η Gazprom και οι εταίροι στην αρχή ήθελαν να αναπτύξουν από κοινού σε κοινοπραξία ε, τον αγωγό αυτό. Όλες αυτές οι εταιρείες ε, και παράγουν και διαθέτουν φυσικό αέριο. Αλλά από ό,τι φαίνεται η Gazprom ε, θα κατασκευάσει τον αγωγό αυτό μόνη τη. Σύμφωνα με το άρθρο 9.1 τη Οδηγίας για το Φυσικό Αέριο, η νέα η αγωγή και η υποδομή θα πρέπει θα, για να εγκριθεί να είναι αποσυνδεδεμένη από το διαχειριστή. Δηλαδή δεν θα πρέπει ο ίδιος να την κατασκευάζει και να διαθέτει και το αέριο. Ε, είναι ενδιαφέρον ε, πλέον που το αναλαμβάνει μόνη της η Gazprom και έκτοτε η γλώσσα της γερμανικής κυβέρνησης έχει κάπως αλλάξει. Τώρα λέγει η γερμανική κυβέρνηση ότι είναι ιδιωτικό αυτό το έργο ό,τι και να σημαίνει. Ότι είναι τελείως ιδιωτική πρωτοβουλία χωρίς οποιαδήποτε πολιτική στήριξη. Αυτό το βρίσκω λίγο ε, έτσι προβληματικό και οδηγεί σε σύγχυση. Οι Γερμανοί πολιτικοί εξακολουθούν να πιέζουν πάρα πολύ και να ασκούν άγριο λόμπι για το Nord Stream 2. Ορισμένοι, ορισμένοι Γερμανοί πολιτικοί, λέει κάποιος, ναι, ορισμένοι Γερμανοί πολιτικοί και στη διάσκεψη ασφαλείας της Ρήγας το 2016, όπου ο Κρίστιαν Σμιτ, υπουργό Γεωργίας της Γερμανίας, είπε ότι αυτό είναι ένα ιδιωτικό έργο κάπου στο βορρά. Ε, ε, βέβαια αυτό δεν είναι απεγκιστρωμένο από όλη τη συζήτηση γίνεται μια συζήτηση για το ρόλο του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία που φαίνεται να έχει αποσυνδεθεί τελείως από το Nord Stream 2. Αυτό που μόνο του είναι αξιοσημείωτο γιατί είδαμε τι ρόλο παίζει η Gazprom που είναι κρατική εταιρεία. Είναι ενδιαφέρον αυτό που ακούσαμε από κάποιους Γερμανούς εκπροσώπους ότι μας διαβεβαίωσαν ότι μετά το 2019 θα είναι εγγυημένος ο ρόλος ε, του τράζιτ της ε, διαμετακόμισης από την Ουκρανία. Αλλά οι Ρώσοι δεν λένε τα ίδια καθόλου. Ούτε αφήνουν να εννοηθεί κάτι τέτοιο. Πάω σε κάποιες σκέψεις τώρα γεωπολιτικές και ασφαλείας. Θα ήθελα να εστιάσω ιδιαίτερα στο ρόλο που διαδραματίζει εδώ η Σουηδία, κράτος μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Σουηδία δεν ανησυχεί πάρα πολύ για την ίδια της ασφάλεια και τον αναφοδιασμό από τον Nord Stream 2. Αυτό που την ανησυχεί είναι θέματα ασφαλείας με την ε, σκληρή έννοια και την ευρύτερη. Ε, πέρα από τις ε, απτές και χειροπιαστές συνέπειες που θα έχει για την ίδια την επικράτεια της χώρας η κατασκευή του έργου. Γενικότερα, τι λέει η Σουηδική κυβέρνηση στις εκτιμήσεις που κάνει. Θεωρεί τη Ρωσία ως μια χώρα που μπορεί να απειλήσει την ε, Βαλτική θάλασσα και άλλες χώρες στρατιωτικά. Η Σουηδία που δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ έχει πολλούς λόγους να ανησυχεί και να φοβάται. Υπάρχει ένα παράδειγμα που μας βοηθάει να το καταλάβουμε. Η Σουηδική επικράτεια είναι στρατηγική σημασία για το ρωσικό στρατό και αυτό επιβεβαιώνεται από διάφορα κατασκοπευτικά πλοία ε, που ε, κατασκοπεύουν και το έδαφος της Σουηδίας ε, και μάλιστα παρατηρούν το νησί Γκότλαντ και τι κάνει και ο Σουηδικός στρατός και οι θελοντές της φρουράς της Σουηδικής. Και επίσης Ρώσοι πράκτορες που υποθέτει τους τουρίστες πάνε εκεί στο νησί της Γκοτλάνδη και κάνουν διάφορες ερωτήσεις σε στρατιωτικό προσωπικό, ε, σε διάφορους εθνοφρουρούς, τι κάνετε εδώ, ποια είναι η δουλειά σας κτλ. Αυτές οι δραστηριότητες έχουν ενταθεί από τότε που ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Σουηδίας ε, πήρε την απόφαση να εγκατασταθεί μόνιμη στρατιωτική παρουσία στη Γοτλανδία έξι μήνες πριν ε, τον προγραμματισμό. Ε, υπάρχει ένα θέμα ότι ε, θα πρέπει να δοθεί ένα λιμάνι σε αυτό το νησί για τον αγωγό ε, και οι Σουηδοί αντιδρούν και ένα δημοτικό συμβούλιο σε μια πόλη που στο παρελθόν είχαν προγραμματίσει να αφήσουν τον Όστριμ να χρησιμοποιήσει το λιμάνι τους έχουν αναστείλει την απόφαση αυτή και ε, ε, το Δημοτικό Συμβούλιο και ο Δήμαρχο πάνε στη Οχόλμη για να συζητήσουν αυτό το θέμα. Και από ό,τι άκουσα σήμερα το πρωί, παρόλο που ανησυχεί η Σουηδική κυβέρνηση και επανειλημμένα το έχει εκφράσει, ε, ε το θέτει αυτό υπόψη των αρχών της τοπικής αυτοδιοίκησης στο Κάσχομ, αλλά από ό,τι φαίνεται πρόκειται να αφήσουν την Κάσπρομ να κατασκευάσει εκεί τις υποδομές. Υπάρχουν λοιπόν ε, συνακροάσεις, υποκλοπές, ε, κατασκοπευτικές ενέργειες και αυτό είναι ενδεικτικό του γεγονότος ότι η ίδια η Σουηδική κυβέρνηση έχει καταλάβει ότι υπάρχουν θέματα ασφαλείας εκεί. Ε, ίσως και να το ανέμεναν. Τώρα, θα πρέπει να τονίσουμε το εξής. Όταν κατασκευάζονται διάφορες υποδομές, βλέπε σύνδεση ηλεκτρική ε, Nordbalt, Σουηδίας, Λιθουανίας. Τι έγινε όταν χτιζόταν αυτή η γραμμή. Είχαν αντισταθεί πάρα πολύ οι Ρώσοι με την παρουσία του ρωσικού στόλου της Βαλτικής θάλασσας για να ε, αποτρέψουν τη δημιουργία αυτής της σύνδεσης. Αυτό δεν ήταν μόνο περιφρόνηση για την εθνική κυριαρχία και την επικράτεια της Λιθουανίας, αλλά ήταν και ένα ε, σημείο ότι θεωρεί την ε, αποκλειστική ζώνη ελευθέρων συναλλαγών της Λιθουανίας ως δικό της χώρο και επικράτη ακόμα η Ρωσία. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον εμπορικό ρόλο του αγωγού αυτού, αν δούμε όλη τη σύνδεση, ε, ξέρετε το Καλίνιγκρατ δεν χρησιμοποιούνται οι λιμενικές εγκαταστάσεις. Για ποιο λόγο αυτό εμπορικά. Αν δούμε ε, ότι το κόστος και το εργασιακό και της αποθήκευσης είναι πολύ χαμηλότερο στο Καλίνιγκρατ. Για ποιο λόγο να πάει να γίνει στη Σουηδία. Και αυτό εντάσσεται και στην ευρύτερη προσπαθή του σχεδιασμό της ε, ρωσικής ε, κυβέρνησης να προωθεί την εχώρια αγορά κτλ. Νέους εμπορικού θα είχε νόημα λοιπόν να χρησιμοποιηθεί ως λιμάνι το Καλίνιγκρατ. Για ποιο λόγο λοιπόν, να το δεις από αμυγός εμπορική σκοπιά αυτό. Έρχομαι τώρα στη Γερμανία. Η Γερμανία θεωρεί το Nord Stream 2 ένα τρόπο να λύσει τα ουσιαστικά προβλήματα που έχει στην προμήθεια φυσικού αερίου. Ορισμένοι πάλι στη Γερμανία, εντάξει. Αφού πήρε την απόφαση να γίνει αυτή η ενεργειακή αλλαγή και να φύγει από τα πυρηνικά. Τελείως. Ορισμένοι λοιπόν ε, Γερμανοί βουλευτές θεωρούν αδιανόητο η Ρωσία να χρησιμοποιεί ε, τους φυσικούς, φυσικού αερίου ως εργαλείο ε, γεωπολιτικής και γεωστρατηγικής. Αλλά δεν σημαίνει ότι αυτό είναι αδιανόητο επειδή δεν έχει συμβεί ποτέ στο παρελθόν το Βερολίνο. Έχει ε, αναλάβει ηγετική θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τη Ρωσία για διάφορες πολιτικές. Ε, αυτό είναι πιθανό να το ξέρει και το Κρεμλίνο στους υπολογισμούς και τους σχεδιασμούς. Και θα κάνει και διαβήματα στην επόμενη γερμανική κυβέρνηση να έρθουν οι κυρώσει τη Ευρωπαϊκής Ένωση προ τη Ρωσία και άλλα. Και αφού η ε, Γερμανία θα είναι κομβική ε, στο μέλλον και για την παρουσία του ΝΑΤΟ στη Λιθουανία, η ε, Ρωσία προσπαθεί να αξιοποιήσει κάθε δυνατότητα που έχει και κάθε μοχλό που έχει να εκμεταλλευτεί για να πιέσει τη Γερμανία προς το δικό της όφελος. Και τώρα, τελειώνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ λίγο ε, στην ε, ευρύτερη γεωστρατηγική εικόνα και το παιχνίδι που παίζετε εδώ. Ε, κοιτάξτε τι γίνεται στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και εδώ διαφωνώ με την εκτίμηση του συναδέλφου Προλαΐσαντος. Ε, αν δείτε λοιπόν τη διαπραγματευτική θέση και τη δυνατότητα πίεσης που έχουν ορισμένες χώρες διαμετακόμισης, με το North Stream 2 λένε ότι εκτίθεται περισσότερο χώρες όπως η Πολωνία, η Σλοβακία και η Ουκρανία και ότι η διαπραγματευτική τους ε, δύναμη απέναντι στη Ρωσία θα μειωθεί. Αν δούμε όμως την ευρύτερη εικόνα, όχι μόνο τον αγωγό Nord Stream 2, αλλά και την κατασκευή του τουρκικού αγωγού φυσικού αερίου, έχει ενδιαφέρον να δούμε εδώ τι συμβαίνει. Και αν δείτε ε, ποια είναι τα σχέδια της Τουρκίας, θα είναι διπλός ο αγωγός 50 με 75 BCM. Το πρώτος θα ε, αντικαταστήσει τον αγωγό που περνάει τώρα από Ουκρανία, Ρουμανία ε, μέσω Μολδαβίας. Δεν έχουμε ε, περισσότερες ποσότητες φυσικού αερίου. Αυξάνεται εκεί η ζήτηση. Από πλευράς εμπορικής έχει νόημα να κατασκευαστεί αγωγός προς την Τουρκία. Γιατί δεν το έκαναν η Ρωσική Ομοσπονδία και η Gazprom προηγουμένως με το South Stream. Και έκανα το South Stream που δεν ήταν αρκετά μεγάλη η ε, ζήτηση στην Ευρώπη. Λοιπόν, η Τουρκία δεν χρειάζεται όλο αυτό ε, δηλαδή 50 με 75 BCM ε, δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα, αλλά θα υπάρχει πλεόνασμα ας πούμε, 8 BCM, ότι θα είναι το πλεόνασμα. Και πού θα πάει αυτό το φυσικό αέριο. Στην νοτιοανατολική Ευρώπη, στην Ελλάδα, σε άλλες χώρες της Βαλκανικής. Αυτό δεν είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον για την Gazprom, δεν είναι βασική της αγορά. Η Γερμανία είναι η μεγαλύτερη και δεύτερη είναι η Ιταλία. Δηλαδή, σημαντικός πελάτης και τελικός προορισμός για την Gazprom είναι η Ιταλία. Το θέμα είναι πώς θα φτάσεις εκεί, θα φτιάξεις νέο αγωγό από αυτή την περιοχή που τελικά θα πρέπει να μοιράζεσαι που ε, είναι στο τρίτο πακέτο το ενεργειακό. Αυτό είναι πολύ απίθανο. Αν δούμε τι έχει κάνει στο παρελθόν η Gazprom, δεν προτιμάει τέτοιες δράσεις. Αυτό που μάλλον θα κάνουν είναι να θελήσουν ε, από τον ITGI που είναι ε, Τουρκία, Ελλάδα, Ιταλία να χρησιμοποιήσει ε, κάποια δυνατότητα, κάποια χωρητικότητα και αν επεκταθεί αυτός ο αγωγός με άλλους θα δημιουργήσει μία οδό προς την Ιταλία που εξαιρείται από τις απαιτήσεις TPA για 25 χρόνια. Υπάρχει και το τάπο από το Αζερβαϊτζάν, Ανδριάτη, μπορεί ε, στο μέλλον να φτάσει τα 20 BCM και παραπάνω. Λοιπόν, εδώ υπάρχει μια διελκυστίδα, ένα παιχνίδι. Ποιος θα φτάσει πρώτο στην Ιταλία, το Αζερβαϊτζάν ή οι Ρώσοι. Είναι ένας ανταγωνισμός και δεν ξέρω κάποια στιγμή μπορεί να είναι και το Ιράν με το πετρέλαιο και άλλοι. Αυτή είναι μάλλον η στρατηγική που ε, ακολουθεί στην Ανατολική η ε, Ευρώπη, η Γκάσπρομ ε, προσπαθεί να φτάσει πρώτη στην Ιταλία. Τέλος, θα ήθελα να πω ότι από τη σκοπιά της Ενεργειακής Ένωσης είναι πάρα πολύ λίγα τα σημεία με τα οποία συμμορφώνεται ο γογός Nord Stream 2. Αλλά κάτι άλλο που έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία είναι ότι αν η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίξει το Nord Stream 2 θα σημαίνει ότι ε, το μοντέλο της ε, Gazprom ή είδε πόσο θέση που έχει στην εγχώρια αγορά αυξάνεται. Ενώ τώρα αυξάνονται οι πιέσει από άλλε εταιρείε όπως είναι η Novatec και τα λοιπά. Λοιπόν, στην εγχώρια αγορά η Gazprom πιέζεται και ποντάρει σε αυτές τις μεγάλες επενδύσεις, τα μεγάλα έργα ε, προς την Ευρώπη. Η, αν το επιτύχει, θα μειωθεί η, πίεση, που έχει και στην εγχώρια αγορά για να σπάσει το μονοπόλιο τη. Και αν η Ευρώπη θέλει ανταγωνισμό, ε, δεν θα πρέπει να ε, δημιουργήσει ένα σενάριο που θα βρεθεί εγκλωβισμένη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ που τηρήσατε ακριβώς το χρόνο σας. Θα ακούσουμε τώρα την κυρία ε, Λόσκο Χότα παρακαλώ, ένα τέταρτο παρακαλώ. Okay. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Θα ήθελα να σας δείξω και διαφάνειες με την ε, παρουσίασή μου. Να σας πω βεβαίως ότι είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ. Να μιλήσω κι εγώ για τον Nord Stream 2 ε, μερικά θέματα ήδη αναφέρθηκαν και επομένως δεν υπάρχει λόγος να δείξω όλα ε, τα, ε, τις διαφάνειές μου. Έχουμε ήδη μιλήσει για το πώς ξεκίνησε, από πού περνάει κτλ οι προκλήσεις ε, είναι σημαντικές, σημαντικότερη εκ των οποίων ε, είναι η απόφαση για το κατά πόσο χρειάζεται μια νέα μορφή συνεργασίας ανάμεσα ε, στην Gazprom και τους Ευρωπαίους εταίρους ε, και οι δυνατότητες χρηματοδότησης ε, του έργου. Αλλά βεβαίως ε, η κυριότερα πρόκληση αφορά το νομοθετικό πλαίσιο και τον δρόμο με τον, οποίο αυτό εφαρμόζεται στο Nord Stream και τον τρόπο με τον οποίο αυτό το σχέδιο θα έχει επιπτώσεις στην Ευρώπη. Ξέρετε ότι έχουν προκύψει και ρυθμιστικά και περιβαλλοντικά ζητήματα, αλλά κυρίως λαμβάνοντας υπόψη το πολιτικό περιβάλλον έχουν προκύψει και πολιτικά ε, προβλήματα και πολιτικά ζητήματα. Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι υπάρχει αυτή η ενδυνάμωση της αντιπαράθεσης Ρωσίας-Ουκρανίας. Έχουμε επίσης ένταση σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσίας, αυξημένες προκλήσεις ασφάλειας. Τα ακούσαμε για τη Βαλτική θάλασσα από τους προηγούμενους συναδέλφους. Αυτό που είναι σημαντικό κατά τη δική μου άποψη είναι να δούμε τις εσωτερικές προκλήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, ας πούμε το Brexit είναι μια από τις κύριες ε, προκλήσεις κατά αυτήν την έννοια. Θα πρέπει να δούμε ποιος μπορεί να είναι ο αντίκτυπος αυτού του Nord Stream. Βλέπουμε ότι ο αντίκτυπος ε, ε, ήδη έχει αρχίσει στην Ευρώπη αυξάνει ας πούμε τις αντιπαραθέσεις σε γενικές ε, γραμμές ε, είναι δύο οι διαφορετικές απόψεις. Η μία εκπροσωπείται από αυτούς που θέλουν το Nord Stream και ε, θα ήθελα εδώ να βασιστώ και σε αυτά που είπαν και οι συνάδελφοί μου. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι θεωρούν ότι το σχέδιο αυτό είναι εμπορικό ε, και επομένως μακροπρόθεσμα ε, θα ε, μειώσει, θα βοηθήσει στις μειώσεις των εισαγωγών φυσικού αερίου. Λένε επίσης ότι θα προκύψει σταθερότητα και ασφάλεια των προμηθειών και μάλιστα με χαμηλότερο κόστος και επίσης ότι η συνεργασία με την Ρωσία μπορεί να οδηγήσει σε συγκεκριμένα οικονομικά ωφέλη τους εμπλεκομένους. Ε, επίσης, ε, αυτή η ομάδα όσον αφορά τις ε, σχέσεις με την Ρωσία επιδιώκει την εξομάλυνση ή την de facto ενίσχυση των σχέσεων και όσον αφορά τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρεί ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερη αναμεξη Επίσης υπάρχει άλλη ομάδα η οποία θεωρεί ότι αυτό το project είναι πιο πολύ πολιτική ε, ε, ότι η οποιαδήποτε ε, εξασφάλιση της προμήθειας θα είναι μονάχα μέσο και βράχη πρόθεσμη και μπορούν να προκύψουν σοβαροί κίνδυνοι διακοπής και επίσης ανάλογα με την θέση της Ρωσίας θεωρούν ότι αντιθέτως μπορεί να αυξήσει την ανασφάλεια, μπορεί να προκύψει αύξηση τιμών κυρίως εάν η Gazprom βρεθεί σε δεσπόζουσα θέση στην αγορά ε, και ότι ναι θα, υπάρχουν, θα υπάρξουν οπωσδήποτε επιπτώσεις στον τομέα ε, του αερίου αλλά θα υπάρξουν επιπτώσεις και στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας και επομένως ε, θεωρούν ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όσον αφορά τις σχέσεις με τη Ρωσία λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση στην Ουκρανία κλπ. Στο χάρτη αυτό βλέπετε ότι η Ευρώπη είναι μοιρασμένη ε, όσον αφορά το Nord Stream. Με μπλε χρώμα έχω βάλει τις χώρες ε, οι οποίες ε, είναι υπέρ του Nord Stream, με κίτρινο αυτές που είναι κατά. Βλέπετε όμως ότι υπάρχουν και κάποιες χώρες που τις έχω βάλει ριγέ. Αυτές είναι οι χώρες οι οποίες αμφιταλαντεύονται, οι οποίες διστάζουν, βλέπουν κάποια στοιχεία θετικά. Ας πούμε, η τσεχική δημοκρατία ε, θεωρεί ότι μπορούν να υπάρξουν ε, θετικές οικονομικές επιπτώσεις από το Nord Stream, αλλά διαβλέπει επίσης ε, και προκλήσεις σχετικά με την ασφάλεια. Επίσης υπάρχουν και οι χώρες οι οποίες έχουν αποφασίσει να κρατήσουν ουδέτερη θέση λόγω της ευαισθησίας του θέματος. Αυτό που βλέπετε είναι ότι ήδη ο Nord Stream πριν ξεκινήσει ε, ε, μοιράζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προκαλεί σύγχυση ε, και επομένως θα μπορούσε να κάνει την Ευρώπη πιο ασθενή, να εξασθενήσει κατά κάποιο τρόπο την θέση της Ευρώπης. Το θέμα της συζήτησης βεβαίως είναι ε, οι κυριότερες προκλήσεις ε, καθώς και ο κεντρικός στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την ασφάλεια ε, της προμήθειας αερίου. Επίσης θα πρέπει να λάβει υπόψη τους υφιστάμενους δεσμούς ανάμεσα στην οικονομία, την πολιτική και τις αγορές του αερίου. Σε αυτό το τελευταίο στοιχείο έγκυται ε, και το πιο δύσκολο σημείο του Nord Stream 2. Ε, γνωρίζουμε ότι και με από το Nord Stream 1 ότι ο ρόλος της ε, Gazprom είναι ήδη σημαντικός και με το Nord Stream 2 κινδυνεύει να γίνει ακόμα μεγαλύτερος. Το 2016 η Gazprom έδωσε περίπου 10% του ε, αερίου της ε, ε, Γερμανίας και αντιπροσώπευσε το 50% της κατανάλωσης αερίου στην Γερμανία και επομένως με τον τρόπο αυτό ενδεχομένως θα ενδυναμωθεί ακόμα περισσότερο ο ρόλος της Gazprom στην αγορά της Γερμανίας καθώς επίσης και στην αλυσίδα προμήθειας στην Γερμανία και στην περιφερειακή αγορά. το North, ο North Stream ενδεχομένω ε, θα μπορούσε να είναι υπεύθυνο και για, το, για την επιπλέον ε, ε διεύρυνση του μεριδίου ε, του ρωσικού αερίου στις εισαγωγές αερίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ είχαμε αύξηση το 2016 και η ε, Gazprom αύξησε κατά 3% ε, σύμφωνα με πρώτες εκτιμήσεις ε, την, ε, τις, τις της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. επομένως αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ακόμα πιο δεσπόζουσα θέση της Gazprom και σε ακόμα μικρότερες δυνατότητες διαφοροποίησης της προμήθειας αερίου, κυρίως για χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Η επίπτωση στην αγορά μπορεί να είναι πάρα πολύ μεγάλη. Αυτό θα μπορούσε να έχει σαν αποτέλεσμα την ακόμα πιο αυξημένη παρουσία της Gazprom στην, ε, στις ανατολικές ε, χώρες Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης και ενδεχομένως θα μπορούσε ε, να δημιουργήσει προβλήματα στη διαδικασία αντιτράστ που έχει ξεκινήσει ήδη η Κομισιόν εναντίον της ε, Gazprom και ενδεχομένως ε, θα αποσταθεροποιήσει λίγο τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης, οπωσδήποτε, ο Nord Stream 2 θα έχει επιπτώσεις και στις εξωτερικές σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης που σχετίζονται με το αέριο, αλλά όχι μόνο. Ε, αυτή τη ε, ε, στιγμή ο κύριος στόχος της Gazprom είναι να ξεπεράσει την την διέλευση από την Ουκρανία και αυτό σε μέσο και βράχη πρόθεσμο περιθώριο και αυτό θα μπορούσε να τροποποιήσει εντελώς τον χάρτη του αερίου. Ε, ο Nord Stream 2 θα μπορούσε ενδεχομένως ε, να αποδυναμώσει τη θέση της Ουκρανίας και την οικονομική και πολιτική ε, σταθερότητα της επίσης θα μπορούσε να σημάνει μείωση της διαπραγματευτικής δύναμης της Ουκρανίας. Ε, θα μπορούσε επίσης ε, να απομειώσει και το ενδιαφέρον των, ε, των operators της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση για, για μεγαλύτερη συνεργασία με την Ουκρανία στον τομέα του αερίου, διότι θα μείωνε τον αριθμό των παροχών προς την Ευρώπη. Επίσης θα μπορούσε ο Nord Stream 2 να δυναμητήσει την εμπιστοσύνη των σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης Ένωσης ε, και ε, Ουκρανίας. Ε, κατά την άποψή μου, το 2014, ας πούμε, ο ρόλος της ενεργειακής κοινότητας άρχισε να γίνεται σταθερό, καθαρότερος και ενδεχομένως θα μειωθεί ο ρόλος της. Επίσης, ίσως να μειωθεί η σκοπιμότητα και η εκπλήρωση μάλλον των στόχων πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, ο Nord Stream 2 θα μπορούσε να επηρεάσει τις εξωτερικές ε, σχέσεις σχετικές με το αέριο με την ε, Ρωσία. Γνωρίζουμε ότι ήδη από το έτος 2014 υπάρχει ένταση ε, στις πολιτικές σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας. Έχουν υπάρξει σύρες κυρώσεων από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι της Ρωσίας και επίσης έχουμε διαπιστώσει και μια ενισχυμένη πολιτική διαφοροποίησης ε, των πηγών ε, προμήθειας ε, ενέργειας. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι στην ουσία δεν έχουν αλλάξει ή μειωθεί οι εξαγωγές αερίου από την Ρωσία και δεν έχουν αλλάξει και οι στόχοι. Εν συμπεράσματι μπορούμε να πούμε ότι ο Nord Stream 2 θα μπορούσε να δυναμητήσει ε, με την ε, δυνατότητα υλοποίησης ορισμένων στόχων της Ενεργειακής Ένωσης ε, σε σχέση ας πούμε με τη διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας θα μπορούσε να αυξήσει την συνεργασία ανάμεσα στις χώρες Ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκής ε, επίσης μπορεί να αποτελέσει ε, πρόκληση για ε, αυξημένη συνεργασία όπως είπα και προηγουμένως κυρίως όμως θα μπορούσε να αποτελέσει έναυσμα για διαφοροποιημένη πολιτική έναντι της Ρωσίας και τροποποίηση των στόχων σε σχέση με τις σχέσεις με την Ουκρανία. Ε, βεβαίως αυτή τη στιγμή ε, τα περισσότερα ζητήματα σχετίζονται ε, με την Ευρώπη γιατί βλέπουμε ότι μπορεί να προκύψουν πολιτικές επιπτώσεις εσωτερικές στις θέσεις γειτονίας κτλ. Ε, Βεβαίω εδώ προσπαθούμε να βρούμε τον καλύτερο δυνατό και όχι τον ιδεώδη κόσμο, ε, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχουν ε, και αγορές οι οποίες ακόμα είναι ρευστές, ας μην λησμονούμε ότι υπάρχει το Brexit. Υπάρχουν επίσης operators ή πρωταγωνιστές ή εμπλεκόμενοι οι οποίοι λειτουργούν με οπορτουνιστικό τρόπο και όχι πάντα με ορθό πολιτικό. Το θέμα είναι να βρεθούν κοινοί στόχοι ε, όσον αφορά την, ε, και κοινή αντιμετώπιση όσον αφορά τη Ρωσία ε, και την Ουκρανία. Ενδεχομένως εδώ θα ήταν μια καλή ευκαιρία να επαναπροσδιοριστούν οι ορισμοί και οι στόχοι. Ε, και ίσως ήρθε η ώρα να συζητηθεί και το θέμα της ενότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή ε, πώς είναι δυνατόν ε, να εξακολουθήσει η ενότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περιπτώσεις όπως αυτή του Nord Stream 2. Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σαν ένα εργαλείο έτσι ώστε να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη, η συνεργασία και η αλληλεγγύη στην Ευρώπη. Θα μπορούσε να αποτελέσει μια καλή ευκαιρία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, λέει ο Πρόεδρος, τους τρεις ε, και τώρα θα ξεκινήσει η συζήτηση, έχουμε χρόνο. Ο κύριος Μπαλτσίτης... Ε, Αλλά πριν ο Τούνε Κέλαμ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τους τρεις ομιλητές μας για την ενδιαφέρουσα ε, προσέγγιση τους αλλά δεν θα πρέπει να χάσουμε τη συνολική εικόνα προφθαλμού. Δεν μπορούμε να υποδηθούμε ότι είναι ξεχωριστή ιδιωτική ε, πρωτοβουλία μόνο ο αγωγός Nord Stream 2. Ακούζοντας τις παρουσιάσεις, είχα την αίσθηση ότι συχνά εμείς οι πολιτικοί δρούμε σαν ε, ε ένας τυφλός που ε, ψηλαφάει ένα ελέφαντα και προσπαθεί να καταλάβει τι είναι. Ε, αποσπασματικά. Εμείς οι πολιτικοί δεν μπορούμε να δούμε αποκομμένα και να εστιάσουμε στα οικονομικά στοιχεία ή στα νομικά στοιχεία. Θα πρέπει να βλέπουμε τη σύνολη εικόνα. Και σας ευχαριστώ κύριε Στραχώτα που αναφερθήκατε σε αυτό. Απευθύνατε την τελική έκκλησή σας ότι χρειαζόμαστε ενότητα και ρεαλιστική προσέγγιση. It was initiated. I... Γιατί πριν από λίγα χρόνια όταν ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια θυμάμαι ένα γερμανό καγκελάριο που το διεκπαιρέωσε αυτό μάλλον το ξεπέρασε πολύ γρήγορα, σου είπε είναι μια ιδιωτική πρωτοβουλία και δεν μπορεί να επέμβει το κράτος. Μα είναι σαφές ότι πρόκειται για την Gazprom που δεκάδες χρόνια είναι το βασικό εργαλείο της ρωσικής εξωτερικής πολιτικής. Αυτό είναι σημαντικό γιατί το βασικό στοιχείο για μας είναι το στοιχείο της ασφάλειας. Η κατάσταση στη Βαλτική θάλασσα έχει γίνει πολύ πιο σκληρή, κυκλοφορεί ο ρωσικός στόλος και προσπαθεί να ελέγξει και το, με το Καλίνιγρα ως βάση του. Και είπατε κι εσείς αυτό ότι όταν προσπάθησε η Λιθουανία να συνδεθεί με τη Σουηδία ε, ε, ηλεκτρική ενέργεια, ε, ένα σχέδιο ανταγωνιστικό και ένα δίκτυο ανταγωνιστικό, τι άσκησαν είχαν πιέσει, κανονικό bullying οι Ρώσοι. Λοιπόν, αυτό ο νέος αγωγό θα αυξήσει το ρόλο, θα αναβαθμίσει το ρόλο της Gazprom και στις γερμανικές και στις ευρωπαϊκές αγορές. Άρα, αυτό που χρειαζόμαστε και έρχομαι στην ερώτησή μου. Βλέπετε καμιά δυνατότητα να εκβιάζει η Ρωσία όχι μόνο για την παροχή φυσικού αερίου, ότι να, κλείνει και τη στρόφιγγα όταν έχουμε πολιτικές ή στρατιωτικές ε, κρίσεις. συμφωνώ απολύτως με το βασικό μήνυμα που λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται ε, πολύ πιο ρεαλιστική προσέγγιση, ενότητα και συντονισμό ε, στην αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. Ευχαριστώ κύριε Βαλτσίτης. E, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ είμαι από τη Λιθουανία που αναφέρθηκε σήμερα ε, σε σχέση με τον αγωγό αυτό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εμπειρογνώμονές μας, ε, αλλά εξέτασαν ε, αυτό το θέμα του αγωγού φυσικού αερίου με τρόπο και αντικρουόμενο και αντιφατικό. Εγώ είμαι μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο τα τελευταία 7 χρόνια και έχω ασχοληθεί πολύ εντατικά με το συγκεκριμένο ζήτημα. Ανακύπτει λοιπόν το εξή ερώτημα. Τι καταφέραμε όλα αυτά τα χρόνια. Πρώτος στόχος μας ήταν ευθύ εξ αρχής, από την κρίση της Ουκρανίας και μετά, να μειώσουμε την ενεργειακή μας εξάρτηση. Όλοι καταλάβαμε σαφέστατα ότι το σημαντικότερο στοιχείο ασφαλείας ήταν να έχουμε μία διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και να απαγκιστρωθούμε, να απεξαρτηθούμε από την Ρωσία. Και σήμερα ακούμε ότι καλά δεν είναι και τίποτα τραγικό ε, αυτό το έργο, φέρνει ανταγωνισμό, πέφτουν οι τιμές, είναι οικονομικό έργο. Δεν συμφωνώ καθόλου. Η Λιθουανία έχει μακρά πείρα σε αυτά τα θέματα και επί μία εξαετία πληρώσαμε 30% υψηλότερες τιμές στη Ρωσία για την ενέργεια, διότι ήθελα να μας τιμωρήσει πολιτικά η Ρωσία. Το έτος 2000 είχαμε ε, ένα αγωγό πετρελαίου, ντούσπα, που προμήθευε ε, πετρέλαιο στα δηληστήριά μας. Και όταν αρνηθήκαμε να πουλήσουμε ε, την, το δηληστήριο Μάλλον αποφασίσαμε να το πουλήσουμε στην Πολωνία και ε, μας απομόνωσαν οι, οι Ρώσοι. Και στη συνέχεια φτιάξαμε στον Πούτινγκ ένα τερματικό σταθμό ε, για το πετρέλαιο για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε μια στοιχειώδη ανεξαρτησία ενεργειακή. Ε, αυτό οδήγησε ε, σε θυμό οργή της Ρωσίας και μάλιστα και κάποιοι Λιθουανοί αντέδρασαν. Σας λέω, έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στον τομέα αυτό και έχουμε καταλάβει ότι η αγωγή ε, πετρελαίου και φυσικού αερίου είναι εξίσου σημαντική με κάποια πυρηνικά εργοστάσια. Ε, είναι πολύ σημαντικό να είσαι ανεξάρτητος στην ενέργεια για να μπορείς να φροντίζεις ε, και να προμηθεύεις ενέργεια στα νοικοκυριά και στους διάφορους χρήστες. Και η αγωγή φυσικού αερίου είναι πάρα πολύ σημαντική για τη χώρα μας, επαναλαμβάνω. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να Αντικαταστήσεις το φυσικό αέριο με κάποια άλλη πηγή ενέργειας. Πρέπει να αλλάξει ολόκληρο το σύστημα το ενεργειακό και τροφοδοσίας και προμήθειας. Εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να σταθμίσουμε πάρα πολύ προσεκτικά τα υπέρ και τα κατά. Θα πρέπει να καταλάβουμε τι σημαίνει η πολωνική απόρριψη ήταν πάρα πολύ τεκμηριωμένη και δικαιολογημένη. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή η Ρωσία για να δούμε στο μέλλον πώς θα διαμορφώσουμε την πολιτική μας. Η κυρία Φωτίγκα. Thank you, Chair. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ συμμερίζομαι βεβαίως της, την αρχή της πολωνικής αρχής ανταγωνισμού, οπότε δεν θα αναφερθώ τα επιχειρήματα που έχουν να κάνουν με τον ανταγωνισμό, θα επικεντρωθώ στα ζητήματα τα πολιτικά και στα ζητήματα ασφαλείας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και πριν ξεκινήσει η κατασκευή του Nord Stream 1, η έννοια της χρήσης ε, του, της ενέργειας, του εργαλείου της ενέργειας ε, για λόγους εξωτερικής πολιτικής αναφέρεται ρητά σε επίσημα έγγραφα της Ρωσίας. Το 2006 ήδη άκουσα την πρώτη παρουσίαση και θυμήθηκα όταν τότε εργαζόμουν μαζί με τον κύριο Γερζι Μπούζεκ ε, και ε, υπέρ της ε, διασύνδεσης μεταξύ των νορβηγικών ε, καταστάσεων αερίου και του Ρόζε και αυτό στη συνέχεια υπονομεύθηκε από τις επόμενες κυβερνήσεις και τελικά προωθήθηκε το Nord Stream. Η Πολωνία δεν ήταν αρκετά ισχυρή και οι χώρες της Βαλτικής ήταν νέα κράτη-μέλη, καθώς και η Πολωνία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως ότι εμείς είχαμε κατά νου ένα ευρωπαϊκό project το οποίο τελικά ιτήθηκε από κόνσεπτ τα οποία ενίσχυσαν τη Ρωσία και την εξωτερική της πολιτική εις βάρος των Ευρωπαϊκών. Ήταν προφανές ότι η Ρωσία ήθελε να ε, συντρίψει την ευρύτερη περιοχή, την Ουκρανία, τις χώρες της Βαλτικής αλλά και τη δική μου χώρα. Να τις καταστήσει λιγότερο ανθεκτικές ε, στους εκβιασμούς. Και είχαμε επεισόδια ενεργειακού εκβιασμού. Θυμάμαι επίσης ότι την 1η Σεπτεμβρίου του 2009 Κατά την επίσκεψη του Πούτιν στο Βέστεπλάτε, μπροστά στους δυτικούς εταίρους, μπροστά στην καγκελάριο Μέρκελ, μπροστά σε πολλούς Ευρω... ανατολικοευρωπαίους ηγέτες, ο Πούτιν είπε ότι θα μπορούσε η Πολωνία να ε, συνδεθεί ε, με το ρωσικό σχέδιο εξωτερικής πολιτικής και ο Λες και τότε αρνήθηκε κατηγορηματικά. Και η Ουκρανή υπουργό τότε η κυρία Τιμοσέγκο αποχώρησε από τη συνεδρίαση. Δηλαδή από την αρχή ήταν πολιτικό το ζήτημα. Και τώρα το Nord Stream 2 έρχεται να ε, χειροτερέψει ακόμα περισσότερο, να επιδεινώσει ακόμα περισσότερο την κατάσταση στην περιοχή μου. Επόμενος με ο κύριος Βασικεβίτσιος, παρακαλώ. Ε, Αουστρεβίτσιος, συγγνώμη. Ε, σας ευχαριστώ πολύ ε, που οργανώνετε αυτή την ακρόαση. Θέλω να ευχαριστήσω και όλους όσους πήραν το λόγο ως τώρα. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να αναφερθώ ε, σε μια έκκληση που έρχεται από την Ουκρανία από τις 15 Νοεμβρίου από τη Βερχόβντα Ράνα οι Ουκρανοί συνάδελφοι καθιστούν σαφές να γράφω αυτό ότι η Ουκρανία παραμένει ένας αξιόπιστος εταίρος για τη μεταφορά φυσικού αερίου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν χρειάζεται εναλλακτική οδός ε, τροφοδοσίας. Δεύτερον, κα, κα, ότι το Nord Stream 2 είναι μια επένδυση οικονομικά αδικαιολόγητη που γίνεται σε βάρος του ευρωπαϊκού καταναλωτή και επίσης ε, υπογραμμίζουν ότι αυτές, αυτή η, οι αγωγοί οι οποίοι θα παρακάψουν την Ουκρανία και η κατασκευή του είναι πολιτικής ε, προέλευσης. Ο κ. Πούτιν και πριν από πολλά χρόνια είχε πει ε, περήφανα μέχρι το 2019 ε, η Ουκρανία δεν θα είναι πια χώρα διαμετακόμιση για το ρωσικό φυσικό αέριο. Το χειρότερο είναι ότι τελικά η Ευρώπη γίνεται εταίρος του Πούτιν εδώ. αυτό που δεν πέτυχε το Nord Stream 1 θα το πετύχει το, το 2. Είναι ένα project φωνιάς. Σκοτώνει τους κανόνες ανταγωνισμού της Ένωσης, σκοτώνει την αλληλεγγύη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπονομεύει πολλά από αυτά πάνω στα οποία χτίστηκε η ιδέα της Ενεργειακής Ένωσης. Όταν τα βλέπουμε όλα αυτά, διαπιστώνουμε ταυτόχρονα ότι υπάρχουν ε, άνθρωποι και Ευρωπαίοι πολιτικοί οι οποίοι βρίσκονται πίσω από αυτό το project και είναι πραγματικά ντροπή για τον κύριο Σρέντερ. Ε, αυτός, αυτός ο στρέντερισμός αρχίζει να ε, διαχέεται. Υπάρχουν πολιτικοί οι οποίοι πληρώνονται από την Κάσπρο. πληρώνονται από μια ρωσική κρατική εταιρεία ε, για να δρουν εις βάρος της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Ε, και πρέπει να λέμε ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Διότι δεν δουλεύουν για την Ευρώπη, δουλεύουν για την τσέπη τους και για τον Πούτιν. Ε, αν δούμε τι γίνεται με τις κρατικές εταιρείες, τα διοικητικά συμβούλια, ε, της Κάσπρομ, ποιοι είναι επικεφαλής. Είναι πρώην μέλη της ΚΑΓΕΜΠΕ. Είναι πολιτικό το σχέδιο, προφανώς. Λοιπόν, τι πρέπει να γίνει από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης για να προχωρήσουμε ε, στην, πρέπει να αξιολογήσουμε τη συμμόρφωση με τους κανόνες ανταγωνισμού της Ένωσης. Ε, πώς μπορεί να ξεκινήσει ένα τέτοιο project χωρίς να υπάρξει αξιολόγηση αντικτύπου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτά σας ευχαριστώ για την ανοχή σας, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ήσασταν σαφείς. Thanks. I would like uh, to start with... Ευχαριστώ. Θα ήθελα να αρχίσω με ένα σχόλιο, ε, όπως και ο κύριος De Jong. Εκτός συζήτησης, όλο το σχέδιο ε, και το έργο αυτό έχει να κάνει με την υλοποίηση της Συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, σέβεται αυτή τη συμφωνία, την ε, πρεσβεύει ή παίρνει ήδη αποστάσεις. Γιατί έχουμε ένα γιγαντίο έργο τώρα υποδομής και περισσότερο όχι μόνο ένα. Λοιπόν, του, του λεχθέντος θα ήθελα να επανέλθω λίγο στη συζήτηση για θέματα ασφαλείας που συνδέονται με τη στρατηγική της Gazprom. Συμφωνώ με ορισμένους ε, συναδέλφους που ήδη τοποθετήθηκαν. Τίποτα δεν μας κάνει να πιστεύουμε ότι αυτό το έργο της Gazprom είναι δώρο προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί πριν από λίγο χρόνο διάβασα ένα άρθρο όπου φερόταν ο κύριος Μετβιέτεφ να λέει ότι θα σας κάνουμε δώρο αυτή την υποδομή φυσικού αερίου και θα σας βοηθήσει η Ρωσία και η Γκάσπρομ για το ενεργειακό μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι εξασφαλισμένο. Ούτε δευτερόλεπτο δεν θα ε, πιστεύω αυτά. Αν δει κανεί ποια είναι η εξωτερική ε, δράση και δραστηριότητες της Ρωσίας εδώ και κάποιο καιρό. Και ποια είναι η απάντηση, τουλάχιστον εν μέρη, απέναντι στις προκλήσεις του Πούτιν και της Ρωσίας, είναι η Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση. Όλο για και περισσότερο για μένα όμως, το έργο αυτό, Nord Stream 2 και άλλη μεγάλη αγωγή, ε, συγκρούονται με τις βασικές ιδέες μας για περισσότερη διαφοροποίηση και λιγότερη εξάρτηση και περισσότερη ενεργειακή ασφάλεια για την Ευρωπαϊκή Ένωση. σε αυτό αποσκοπεί η μεγάλη ιδέα της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Ένωσης. Και τίθεται το ερώτημα, εμείς ως Ευρωπαίοι και Ευρωπαίοι πολιτικοί, όχι μόνο εδώ, γενικότερα, και μιλώ και για τους ε, εθνικούς συναδέλφους. Θα μπορέσουμε να αντιταχθούμε σε αυτές τις συγκρούσεις ε, για να έχουμε μεγαλύτερη ομόνοια ε, για την δική μας ενεργειακή ένωση. Έχει πολύ μεγάλη σημασία και για την ίδια την Ουκρανία αλλά και για μας. Και τέλος, επειδή δεν θέλω πάντα να βλέπουμε τους Ουκρανούς ε, ως κάποιους που μας ζητάνε ε, συνέχεια κάποια πράγματα. Η μεταρρύθμιση της Λαφτογκάς, της Ουκρανικής, είναι από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα αυτό τον καιρό και κατάφερε η Ουκρανία να μειώσει την κατανάλωση του φυσικού της αερίου και αυτό είναι καλό ε, μήνυμα ότι δεν ε, έρχονται συνέχεια σε εμά για να μας ζητούν διάφορα πράγματα, αλλά συμμετέχουν και ανταποκρίνονται στις διάφορες προκλήσεις ενεργειακέ. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε ακόμα τρεις εγγεγραμμένους ομιλητές. Γκάλερ, Γιούρεκ και Κόβεν Μίκερ. Ο κύριος Κόβεν Μίκερ πρώτος. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συζητάμε τώρα για την επίπτωση του Nord Stream σε ευρωπαϊκές χώρες, χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλάμε για τις πολιτικές συνέπειες, μιλάμε για την τύχη της Ουκρανίας, αλλά κανένας δεν συζητάει μια χώρα ε, που είναι η Ρωσία και η οποία, στην οποία έχει η επίπτωση. Ο Λουκασέγκο προσπάθησε να Eh, ε, συγγνώμη για την Ρωσία. Ε, ο Λουκασέγκο προσπάθησε να αναφερθεί στο θέμα αυτό και ε, ε, είναι αλήθεια ότι το χρησιμοποιεί και σαν σαν μοχλό πίεσης και βεβαίως η Ρωσία πολύ θα ήθελε να έχει μοχλοπίεσης και ε, απειλής ε, προς τον κύριο Λουκασένκα. Είναι γνωστά τα αισθήματά μου βέβαια για την ε, Ρωσία, αλλά παρόλα αυτά το ζήτημα της Λευκορωσίας θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Ο Μιχαήλ Γκάλερ. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι τα περισσότερα έχουν ήδη υποθεί. Έχω όμως ένα προβληματάκι. Δηλαδή, ε, εγώ συμμερίζομαι τα τρία ευρήματα σας, αλλά νομίζω ότι ε, θα έπρεπε να έχουμε και κάποιον εκπρόσωπο της Γκάσπρομ ή τέλος πάντων κάποιον από την άλλη πλευρά, ε, από την Πάσφα, από οποιονδήποτε. για να ακούσουμε και τα δικά τους ε, επιχειρήματα. Έχουμε εδώ εμπειρογνώμονες οι οποίοι έχουν μια διαφορετική άποψη. Πάντως, νομίζω ότι είναι σαφές ότι όλοι θέλουμε διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας. Επίσης, θέλουμε μια, ε, έναν ικανοποιητικό όγκο, ε, έτσι ώστε να έχουμε δυνατότητα να πέσουν, τις, να πέσουν οι τιμές. Η ερώτησή μου ε, είναι διτή σχετικά με τον Nord Stream 2 ε, όλη αυτή ε, η όλες αυτές οι χώρες από τις οποίες περνάει θα μπορούσαν ενδεχομένως να κάνουν μια επιπλέον μελέτη περιβαλλοντικού αντικτύπου ε, αλλά βεβαίως ε, ενδεχομένως ε, θα μπορούσε με τον τρόπο αυτό και να επιμηκυνθεί ο χρόνος αλλά και να γίνει πιο ακριβό το σχέδιο αυτό. Εν πάση περιπτώσει όμως θεωρούμε ότι θα πρέπει να προσέξουμε έτσι ώστε οι αποδέκτες να είναι αυτοί οι οποίοι έχουν ανάγκη. Δηλαδή ε, όταν ε, οι διασυνδέσεις ε, είναι περισσότερες και καλύτερες από τη δική μας πλευρά, μειώνεται η δυνατότητα ελέγχου της Ρωσίας. Και ε, βέβαια μπορούν ε, να κάνουν κάποιες ε, παρακάμψεις, αλλά όχι όσον αφορά την τελική κατάληξη. Εγώ θέλω να πω σαφές, όπως, σαφώς, όπως ανέφερε και η, αναφέρθηκε και προηγουμένως, υπάρχει και στην Γερμανία έτσι, διαφοροποιημένη αντιμετώπιση. Ο κύριος Σόλτερ και οι φίλοι του, Σρέντερ και οι φίλοι του έχουν διαφορετική ε, άποψη ε, και το επομένως το θέμα είναι εάν θα, εάν θα θεωρηθεί ε, ιδιωτικό ζήτημα, ιδιωτική επένδυση, ενώ όλοι γνωρίζουν και γνωρίζουμε τι ακριβώς αντιπροσωπεύει η Gazprom. Σε αυτή την περίπτωση απλώς οι οικονομικές θεωρήσεις θα υπερίσχυαν. Ε, νομίζω ότι τέτοιου είδους projects καλό είναι να μην προχωράνε γιατί διαφορετικά η ρωσική επιρροή θα είναι ακόμα περισσότερο. Εγώ σαν δημοκράτη, λέει ο Πρόεδρος, ε, μπορώ να συμφωνήσω με αυτά που λες. Ευχαριστώ. Είναι μια παράδοξη ε, υπόθεση αυτή τώρα, ένα παράξενο έργο. Ακούμε στην Ευρώπη ξανά και ξανά ε, ότι είμαστε κατά του εθνικισμού και του λαϊκισμού. Μα το Nord Stream 2 είναι μνημείο ε, εθνικού εγωισμού η μοίρα μας, η ενεργειακή μας ασφάλεια δεν ενδιαφέρει τη Ρωσία, δεν δίνει δεκάρα. Δεν πρόκειται για την Πολωνία μόνο, πρόκειται και για τις χώρες της Βαλτικής και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας. Αυτούς το μόνο που τους νοιάζει είναι ε, τα οικονομικά συμφέροντα. Δεν υπάρχει ευρύτερη ε, ε, προοπτική. Αυτό είναι κλασική ε, λαϊκιστική τακτική. γιατί σκέφτονται μόνο ε, κοντόφθαλμα μάλιστα το ε, κέρδος. Και επίσης, τι γίνεται με την ανικανότητα των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Ωραία, έχουμε επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία. Οι κυρώσεις αυτές μπορεί να είναι οδυνηρές για κάποιες ελίτ, αλλά δεν πειράζουν καθόλου τη ρωσική στρατηγική και το σχεδιασμό της. Ανέφερε και η κυρία Φωτίγκα τη ε, στρατηγική της Ρωσίας. Θέλουν να επηρεάζουν πολιτικά δια των εξαγωγών. Ε, οι δικές μας λοιπόν ε, κυρώσεις δεν πρόκειται να πλήξουν στρατηγικά καθόλου τη Ρωσία. Εάν δεν σταματήσουμε αυτό το έργο, Nord Stream 2 που εκπροσωπεί αμυγό ρωσικά στρατηγικά συμφέροντα. Βλέπουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι ανίκανη σε πολιτικό επίπεδο. Τα είπε και ο κύριος Γκάλερ προηγουμένως. Εδώ και χρόνια οι Τσέντεου, οι Γερμανοί χριστιανοδημοκράτες, αντιτίθενται σε αυτό το έργο, το οποίο χτίζεται κανονικά. Άρα, πού είναι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη είτε θα σταματήσουμε αυτό το έργο στα πλαίσια των κυρώσεων μας προς τη Ρωσία, είτε θα είμαστε ανήκα να μιλάμε ε, στο μέλλον για αλληλεγγύη. Θα είναι κούφια λόγια και μόνο. Ευχαριστώ κύριε Γιούρεκ. Όλοι οι συνάδελφοι που ζήτησαν το λόγο τον πήραν. Θα έλεγα οι εμπειρογνώμονες να απαντήσουν σε μια σειρά που έγιναν. Ε, θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε ανάποδα αυτή τη στιγμή. Πρώτα οι κυρίες. Ε, έτσι λοιπόν με την αντίστροφη σειρά καλό θα είναι 12 και να ολοκληρωθεί η συζήτηση οπότε έχετε περίπου 5 με 7 λεπτά ο καθένας. Απαντήστε όσο θέλετε, όσο μπορείτε περισσότερε ερωτήσει Σα ευχαριστώ, σα ευχαριστώ και για όλα τα σχόλια και τι ερωτήσει. θυμάμαι δύο άμεσες ερωτήσεις από τον κύριο Γκάλερ. Η μία αφορούσε τις εναλλακτικές που έχουν οι τοπικές αρχές στη Βαλτική θάλασσα για να καθυστερήσουν τον Nord Stream 2. Έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, όντως ε, οι μεγαλύτερες δυνατότητες ε, είναι νομικές. Ε, περνάει από τη Δανία ε, ο αγωγός από τα δανεικά ύδατα η Δανείοι αλλά και άλλες σκανδιναβικές χώρες ε, δεν σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν το αυτονομικό χαρτί αν θέλετε μόνοι τους δεν θέλουν να πολιτικοποιήσουν τη σχέση τους με τη Ρωσία για διάφορους λόγους στην περίπτωση της Δανίας, αν δεν κάνω λάθο και διορθώστε με, αν κάνω λάθο. υπάρχουν κάποια κοινά συμφέροντα στην Αρκτική. Ε, τώρα μετά τέθηκε το ερώτημα, αν το Nord Stream 2 κατασκευαστεί, μπορεί να... Ε, να μεταφερθεί αν θέλετε στην, ε, εσωτερική εσωτερική αγορά με τρόπο που ωφελεί για την Ανατολική Κεντρική Ευρώπη. Είναι δύσκολο να απαντηθεί αυτό. Η εμπειρία του το Nord Stream 1 είναι μικρή ε, και μάλιστα εμφανίστηκε στην τιμή που έπεφταν, στη στιγμή που έπεφταν οι τιμές ε, γενικότερα στα μακροπρόθεσμα συμβόλαια. Μετά υπήρξε μεγάλη ζήτηση από την Ουκρανική πλευρά και αυτό ε, έδωσε έτσι μια όθηση στις ροές μεταξύ Ανατολής και Δύσης, οπότε δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς ποιος ήταν ο αντίκτυπος της Nord Stream 1 ε, υπό κανονικές συνθήκες για να ξέρουμε και τι θα γίνει με το Nord Stream 2. Αυτό μπορώ να σας πω, ποιες είναι, αυτό μπορώ να σας πω εγώ είναι ποιες είναι οι ανησυχίες. Οι ανησυχίες από, στην, στην κεντρική Ευρώπη είναι ότι τα interconnectors, αυτά τα στοιχεία διασύνδεσης που θέλουν να οδηγήσουν στη διαφοροποίηση, και όταν το διαφοροποίηση δεν ο μόνο ανταγωνισμό μεταξύ ρωσικών, ε, δύο, ρωσικών ε, ε, πηγών φυσικού αερίου, Είναι το, ο κίνδυνος λοιπόν να ε, πλημμυρίσουν από ρωσικό φυσικό αέριο. Ε, επίσης ε, μπορεί να μην δημιουργηθούν νέες υποδομές και κατά κάποιο τρόπο αυτό θα μπορούσε να βλάψει τον ανταγωνισμό μακροπρόθεσμα. Λόγω αυτού, αυτό που χρειαζόμαστε πιστεύω είναι μια μελέτη αντικτύπου σε βάθος ε, σε ό,τι αφορά το ποιες θα είναι οι επιπτώσεις για τον ανταγωνισμό, ε, για τη διαφοροποίηση στην κεντρική και στη κεντρική ανατολική Ευρώπη. Και ποιος θα είναι ο αντίκτυπος ε, ε, στην αυξημένη πρόσβαση απευθείας παραγωγών στην τελική αγορά. Και επίσης μια σε βάθος ανάλυση, όπως είπε νωρίτερα πως πως ο κ. Πληθουανία προηγουμένως, ε, μια ανάλυση της πρώτερης εμπειρίας. Όταν δηλαδή το ρωσικό φυσικό αέριο, οι ρωσικές επενδύσεις ε, ενεπλάκησαν με, πολιτικά ζητήματα. Ε, ή όταν είχαμε κάποια διακοπή ανεφοδιασμού που δεν είχε να κάνει ε, με, την, με το πέρασμα από την Ουκρανία. Αυτό χρειάζεται, διότι η συζήτηση για τον Stream 2 προχωράει και θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι μπορεί να οδηγήσει σε βελτίωση των πολιτικών σχέσεων μεταξύ Ρωσία και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, έχουμε όλο και πιο συχνές διμερεί ε, επισκέψεις από τις εταιρείε, ε, προχωράει το Nord Stream 2. Υπάρχει λοιπόν εδώ μια αντίθεση. Αυτά είχα να πω εγώ. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Κύριε Λόσκοτ Στραχώτα. Και τώρα ο κύριος Διόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να απαντήσω στις ερωτήσεις του κυρίου Κέλαμ και του κυρίου Βαλτσίτης. Ε, να απαντήσω μαζί γιατί ήταν επεκαλυπτόμενες οι ερωτήσεις σε κάποιο βαθμό. Ρωτήσατε ε, τι πίεση θα μπορούσε να ασκήσει η Γκάσπρομ στη Γερμανία και η Ρωσία γενικότερα. Δεν χρειάζεται να πάμε πολύ μακριά στην ιστορία για να καταλάβουμε τι πίεση θα μπορούσε να είναι αυτή. Κοιτάξτε τι έγιναν σε χώρες που αντέστρεψαν τη ροή ε, Πολωνία, Σλοβακία και ε, Ουγγαρία ε, προς την Ουκρανία όταν δήλωσε ότι δεν πρόκειται να αγοράσει από την Gazprom ασκήθηκε πολιτική πίεση στις χώρες αυτές και σταμάτησε η Ουγγαρία να προμηθεύει με αντίστροφη ροή αέριο στην Ουκρανία. Ένα παράδειγμα είναι αυτό. Βέβαια, αυτά θα τα δούμε ε, να αυξάνονται εν ώψη σημαντικών αποφάσεων σε ευρωπαϊκά συμβούλια για κυρώσει κτλ. Ε, έχει συμβεί και στο παρελθόν αυτό. Ε, σε σχέση με αυτό που ρώτησε ο κύριος Βαλτσίτης τι κάναμε ε, στην ουσία. Πολλά κάναμε. Ολοκληρώσαμε εσωτερική αγορά ενέργειας με συνθέσεις, Ανάλογα με την πολιτική πίεση που ε, ασκείται, μπορεί ο καθένα να σταματήσει την αντίστροφη ροή, αλλά η δυνατότητα είναι πολύ μεγαλύτερη από το 2009 και αυξάνεται η αντίσταση και έντοχη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Στόχο ήταν να μειωθεί η εξάρτηση. Αν δείτε τι συμφωνήθηκε στην Ενεργειακή Ένωση σε αυτά τα πλαίσια. Αυτό το λέει όλα. Είναι κάπω ε, ε απορίας άξια όταν αντιτίθεται κανείς σε ένα τέτοιο έργο. Αυτά δεν συνάδουν με τα όσα αποφασίστηκαν για την Ενεργική Ένωση. Ε, ο κ. Οστρεβίτσιος τη ρώτησε τι μπορεί να γίνει έτσι ώστε να δούμε κατά πόσο συμμορφώνονται με το δίκαιο ανταγωνισμού. Κοιτάξτε, δεν θα πρέπει να λησμονούμε ότι διέρχεται ο γογός αυτός από χωρικά ύδατα διαφόρων κρατών μελών. Και την τελευταία φορά που το κοίταξα αυτό, στα χωρικά ύδατα των κρατών μελών, ε, ε, ισχύει το κοινοτικό δίκαιο, το ευρωπαϊκό δίκαιο. Και αν δείτε το δίκαιο ε, ανταγωνισμού, και κοιτάξτε ποιος το διαχειρίζεται και ποιος το ε, κατέχει, ποιος είναι ο ιδιοκτήτης, ε, δεν είναι πολύ δύσκολο να δεις αν συμμορφώνεται ή όχι. Αν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να χρησιμοποιήσει διαδικασίες αδειοδότησης ή υπερβελοντικά, εγώ δεν θα πήγαινα σε εκεί. Οι σκανδιναβικές χώρες ε, δεν θέλουν να το πολιτικοποιήσουν, το βλέπουν ως ένα διεθνές ε, ζήτημα και κινούνται βάσει διεθνούς δικαίου. Ε, τώρα, για ποιο λόγο δεν υπάρχει μελέτη αντικτύπου πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής αυτό πραγματικά με ξεπερνάει, δεν το καταλαβαίνω και με εκπλήσει πολύ. Ένα έργο ε, τέτοιου μεγέθους, με τέτοιες συνέπειες, περιβαλλοντικές, πολιτικές, ασφαλείας κτλ. Με αυτό... Ε, είναι προφανέστατο ότι χρειάζεται μελέτη αντικτύπου, όχι επειδή το ζουν διάφορες χώρες. Αυτονόητο, ε, μου φαίνεται. Έρχομαι στην ερώτηση της κυρίας Χάρμς. Συμφωνώ απολύτως ότι η ε, μεταρρύθμιση της ναύταγκας είναι κάτι πολύ σημαντικό και ήδη οι Ουκρανοί έχουν το κλειδί για να λυθεί ε, ε, όλο αυτό το μπέρδεμα. για να δούμε αν έχει νόημα και από το εμπορική σκοπιά. Δεν ξέρω γιατί διστάζουν να το πράξουν οι Ουκρανοί. Είμαστε ακόμα σε θέση, ρωτήσατε, να συμφωνούμε σε θέματα τύπου Ένωση σε ένα πλαίσιο ευρωπαϊκό ε, πέραν δηλαδή των ε, τυχών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σε εθνικό επίπεδο. Θα πρέπει να γίνει μια μελέτη επιπτώσεων ε, για το τι θα σημάνει η κατασκευή ενός τέτοιου αγωγού και καλό θα ήταν να γίνει αυτή η συζήτηση, θα βοηθούσε στη δυνατότητα να ληφθεί σωστή απόφαση για την υλοποίηση της Ενεργειακής Ένωσης. Για λόγους χρονικούς ε, θα σταματήσω εδώ. Ευχαριστώ. Ο επόμενος ομιλητής, ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούν και είναι αναμφισβήτητο γεγονός ότι βεβαίως η ενεργειακή πολιτική είναι οπωσδήποτε ένα, ένα ε, ε, σημείο, ένα τμήμα της ε, πολιτικής και της εξωτερικής πολιτικής της Ρωσίας. Το ζήτημα είναι και το ερώτημα είναι τι μπορεί να κάνει κανείς γι' αυτό. Μια απάντηση που θα μπορούσα να δώσω ήταν πάρα πολύ απλή. Δηλαδή θα μπορούσα να πω μην παίξετε ένα παιχνίδι ε, το οποίο δεν το παίζετε καλά, δηλαδή το γεωπολιτικό ε, παιχνίδι να παίξετε το παιχνίδι το οποίο γνωρίζετε καλά, το οποίο, το οποίο παίζει καλά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, Monkey Game, ε, το οποίο είναι ένα παιχνίδι ε, που θα πιέσει την Gazprom, γιατί η Gazprom χρειάζεται οπωσδήποτε αυτήν την αγορά. Μιλάμε για 178 BCM. Ε, για την Ευρώπη και την Τουρκία. Η Τουρκία ε, επίσης ε, είναι σημαντικό κομμάτι της αγοράς. Τι χρειάζεται την αγορά αυτή η Gazprom οπωσδήποτε. Και αυτό ακριβώς θα πρέπει να χρησιμοποιήσει. Εκεί πρέπει να πατήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. αυτό το ξέρει και το κάνει καλά. Το θέμα των υποδομών, το θέμα των διασυμβέσεων των αγορών την διευκόλυνση επομένων μέσω πολλών σημείων ε, εισόδου ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δυνατότητα πάνω από 2.000 BCM ε, υγροποίησης και επομένως θα πρέπει να χρησιμοποιήσει την αγορά, την δυνατότητα αυτή. Ε, και ε, βεβαίως η Gazprom δεν μπορεί να το αλλάξει αυτό. Δεν μπορεί να αλλάξει το ότι το υγροποιημένο αέριο είναι ε, ο αντίπαλός της. Επομένω, εδώ χρειάζεται να παίξει αυτό το χαρτί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το τελευταίο είναι ε, το λογισμικό. Θα πρέπει οπωσδήποτε να, παίξει ε, καλά, ε, να παίξουν καλά οι κανόνες του ανταγωνισμού και από τη στιγμή που υπάρχουν κανόνες να χτυπήσουν τυπάτε απευθεία στο κεφάλι οποιονδήποτε δεν εφαρμόζει τους ε, κανόνες. Ε, ένα άλλο σημείο βεβαίως είναι, ε, και αυτό είναι απέτηση, θα πρέπει να έχουν όλοι το software, θα πρέπει όλοι να λειτουργήσουν σύμφωνα με τους κανόνες, αλλά αυτό δεν σημαίνει, δεν ισχύει πάντα συχνά στις ανατολικές χώρες. Δηλαδή μέχρι να στηθεί το ρυθμιστικό πλαίσιο, μέχρι να μπουν οι όροι της αγοράς και της, ε, του ανταγωνισμού. Ε, περνάει και ε, καιρός. Θα πρέπει οπωσδήποτε λοιπόν πριν αφήσετε ένα κομμάτι της, της, των δυνατοτήτων σας σε ξένα χέρια να δημιουργήσετε τις υποδομές εσείς οι ίδιοι. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία μου, ευχαριστώ πολύ και τους δύο μας εισηγητές. Ολοκληρώ ολοκληρώθηκε η δημόσια ακρόαση. Ήταν εξαιρετικά καλή ιδέα η οργάνωση αυτής ε, της ε, ακρόασης. Είχαμε μια πολύ καλή συζήτηση ε, σχετικά με τον Nord Stream 2 και τις πολιτικές επιπτώσει Πριν ολοκληρώσω, την, πριν ε, ε, κλείσω την ε, συζήτηση να θυμηθείτε ότι αλλάζουμε αίθουσα. Θα πάμε στο Γιάννα 4-2, 4Q2 στις 3 έτσι ώστε να συζητήσουμε και να ψηφίσουμε για την ευρωπαϊκή πολιτική στην Αρκτική. Ευχαριστώ πολύ για την πρωινή συνεργασία.